Ξαναρχίζουμε κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να απονείμουμε μετάλλιο σε αυτούς που ήρθαν σήμερα το απόγευμα εν Θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή σε μια απόφαση που λάβαμε σήμερα το πρωί για να αναβάλουμε την ε, υποβολή τροπολογιών για την έκθεση ΚΑΝΤΕΚ γιατί δεν έχει γίνει ακριβής μετάφραση σε ορισμένες γλώσσες και αυτή η έκθεση είναι ύψης της σημασίας. Με τη συμφωνία του κυρίου Κάντεκ αναβάλουμε την υποβολή τροπολογιών, την προθεσμία μέχρι τις 11 Μαΐου, δηλαδή την επόμενη Τρίτη. Αλλά η απόφαση αυτή επισύρει και συνέπειες. Και θα ήθελα να σας μιλήσω για την τροποποιημένη θέση η Γραμματεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια σε συνεργασία με την Υπηρεσία Μετάφρασης έτσι ώστε η ψηφοφορία στην Επιτροπή να γίνει στις 2 Ιουνίου όπως είχαμε προγραμματίσει αρχικά. Επειδή όμως την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή το Κοινοβούλιο είναι κλειστό και επειδή η υπηρεσία μετάφραση χρειάζεται 10 εργάσιμες, ίσως ορισμένες μεταφράσεις να φτάσουν στο γραφείο σας μία μέρα πριν από την ψηφοφορία. Να το γνωρίζετε αυτό. Υπάρχει πιθανότητα ότι παρά τις προσπάθειες που θα καταβληθούν μπορεί να μην έχουμε όλες τις μεταφράσεις εγκαίρως για τις 2 Ιουνίου και σε αυτή την περίπτωση θα αναβάλουμε την ψηφοφορία η οποία θα λάβει χώρα στις 22 Ιουνίου στη συνάντησή μας από 9 ε, έως 10 πριν έρθει ο Υπουργός, ο Νορβηγός Υπουργός Αλίας. Άρα θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε η ψηφοφορία στην Ολομέλεια να γίνει τον Ιούλιο. Κάτι το οποίο επιθυμούσε ο κύριος Κάτεκ και τα άλλα μέλη της Επίτροπης. Προσπαθούμε λοιπόν να αρκεστούμε στην απόφαση του πρωινού, αλλά ίσως υπάρξουν δυσκολίες ε, χρονισμού και ίσως η ψηφοφορία γίνει στις 22 Ιουνίου. Αυτό είναι το αρνητικό. Απλώς να το ξέρετε. Αυτή τη βάση θα ακολουθήσουμε. Λοιπόν, ας ξαναρχίσουμε με το θέμα 8 στην ημερήσια διάταξη που είναι ε, ορισμένα είδη υδατοκαλλιέργειας και στόχος για τη χρήση αυτών των ξενικών και απόντων ειδών είναι να λάβουμε υπόψη τον κανονισμό 708 κάθετος 2007 για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξενικών και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών για να αποσύρουμε την γραφειοκρατία με την επαρκή περιβαλλοντική προστασία. Η έκθεση αυτή με συναπόφαση ανατέθηκε στην ομάδα ε, Γκουε, στον κύριο Φερέρα και η απόφαση ε, μάλλον υποβλήθηκε από ε, και εξετάστηκε από την Κομισιόν. Είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και με βάση την, ε, το προσχέδιο κανονισμού που απεστάλλει στις 2 Μαρτίου, ο κύριος Φερέρα θεωρεί ότι θα πρέπει να λάβουν υπόψη μόνο το άρθρα 42.2 σαν την ε, κατάλληλη νομική βάση. δυνάμη του άρθρου 37 του κανονισμού του Κοινοβουλίου, η πρόεδρος κυρία Φράγκα έγραψε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ζητώντας ε, γνωμοδότηση ως προς την καταλληλότητα της νομικής βάσης που προτάθηκε από την Κομισιόν. Η γνωμοδότηση αυτή είναι διαθέσιμη και έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Επίσης, θα ήθελα να σε επισύρω την προσοχή σε μία ε, λεπτομεριακή γνωμοδότηση ως προς την πρόταση, η οποία εγκρίθηκε σε 17 Μαρτίου από την ΟΚΕ και έχει αποστολή ε, για, σε εσά για ενημέρωσή σας. Ο κύριος Φερέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ψηφίσαμε στην Επιτροπή αυτή το πρωί μια σημαντική έκθεση του συναδέλφου Μιλάν για μια στρατηγική εξέλιξης της ε, υδατοκαλλιέργειας. Μία από τις ε, συστάσεις αφορούσε την επιστημονική έρευνα και την τεχνολογικές εξελίξεις ως προς τα αυτόχθονα είδη υδατοκαλλιέργειας. Επίσης υπάρχει η ανάγκη και, υπάρχουν και υπάρχει υποδομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να προωθήσουμε την παραγωγή αυτή την καλλιέργεια αυτών των εξωτικών είδων. Υπάρχει ο κανονισμός της Επιτροπής σε σχέση με τις εγκαταστάσεις με εξωτικά είδη και η Επιτροπή μετά από την πρώτη ανταλλαγή απόψεων εδώ, και με βάση την έκθεση Ίμπας Λάβαμε υπόψη τι επιπτώσει των εξωτικών ειδών στην υδατοκαλλιέργεια. Πρόκειται για μία πρόταση που ορίζει ένα λειτουργικό σχέδιο έτσι ώστε να έχουμε ένα λειτουργικό ορισμό των κλειστών εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας λαμβάνοντας υπόψη και τις ε, τεχνικές προδιαγραφές. Σύμφωνα με αυτό τον ε, ορισμό και με βάση τις οργανώσεις που συμμετείχαν, ο βαθμός κινδύνου θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά, ενδεχομένως σε αποδεκτό επίπεδο, εάν ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διαφύγης των στοχευμένων και μη στοχευμένων οργανισμών. Σύμφωνα με τα καθορισμένα πρωτόκολλα στις εγκατάσταση υποδοχής με βάση τα αποτελέσματα αυτά η Επιτροπή προτείνει την εξαίρεση των εισαγωγών και μεταπτωπίσεων που προϋποθέτουν την χρήση κλειστών εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας έτσι ώστε οι φορείς να μην πρέπει να πληρούν αυτούς τους γραφειοκρατικούς όρους. Στην αιτιολογική σκέψη, η Επιτροπή λέει ότι η εισαγωγή ξενικών ειδών είναι ένας από τους κύριους λόγους ε, κλειδονισμού των οικοσύστημάτων έτσι ώστε να καταστραφούν οι φυσικοί οικότοποι. Και, όπως σημειώνει η Επιτροπή, η εισαγωγή ξενικών ειδών στα ευρωπαϊκά παράκτια και εσωτερικά ύδατα αποτελεί μία από τις πρακτικές υδατοκολιέργειες και πρακτικές που αφορούν την πυκνότητα εκτροφής. Άρα, θα πρέπει να υπάρχει και ένα αντιστάθμισμα. Δηλαδή ένας ορισμός των προαπαιτήσεων σε σχέση με αυτές τις κλειστές εγκαταστάσεις υποδοχής. Καθώς και ένας έλεγχος των εγκαταστάσεων έτσι ώστε να γνωρίζουμε ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι προδιαγραφές. Το ίδιο αφορά και την μεταφορά των στοχοθετημένων ειδών και μη στοχοθετημένων ειδών. Με βάση αυτή την αρχή προτείνουμε μία σειρά από τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής. Ιδιαίτερα 1, 2, 7 έως 13 που όπως ανέφερε ο Πρόεδρος σχετίζονται με προσαρμογές στην θέση σε ισχύ τη συνθήκης της Λισαβόνας, άρα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες αυτών των τροπολογιών. Ζητήθηκε από τον Πρόεδρο μία γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και από τη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου που είναι παρούσα. Ε, αν υπάρχουν αμφιβολίες θα μας διασαφηνίσουν ό,τι θελήσουμε. Και επίσης η γραμματεία πρόθεσε αυτή την εργασία έτσι ώστε να υποβληθούν αυτές οι τροπολογίες. Πρόκειται για την 1, 2 και 7 έως 13 που αφορούν προσαρμογές από θέσεις σε ισχύ της νέας συνθήκης. Υπάρχουν άλλες πέντε τροπολογίες με ένα συγκεκριμένο ε, περιεχόμενο, τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή πέντε τροπολογίες ή περισσότερες βασίζονται σε μια πρόταση του Συμβουλίου και στην γνωμοδότηση που μας εστάλει από την ΟΚΕ. Από την ΕΟΚΕ. Εδώ αναφέρονται διάφορα θέματα που σχετίζονται με το θέμα μας και θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Μία πρώτη, πρώτες του Συμβουλίου με συμφωνία της Κομισιόν εισαγάγει μία προθεσμία που δεν υπάρχει στην πρόταση Επιτροπής. έτσι ώστε να ορίσουμε έναν κατάλογο των κλειστών εγκαταστάσεων στα κράτη-μέλη σε έξι μήνες και υπάρχει και μία διευκρίνηση στον ορισμό της εγκατάστασης, κλειστής εγκατάστασης υδατοκαλλιέργειας που προτείνεται από την ΕΟΚΕ που είναι λογική έτσι ώστε να αρθούν οι αμφισημίες στην εφαρμογή έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη ότι οι κλειστές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας βρίσκονται επί ξηράς όπως ορίζει το έργο Impasse και μία άλλη τροπολογία που διευκρινίζει τις απώλειες ε, υδατοκαλλιέργειας εξαιτίας ε, πλημμυρών, βανδαλισμών, κλοπών έτσι ώστε να υπάρχει μία απόσταση ασφάλειας μεταξύ της εγκατάστασης και των υδάτων. Υπάρχει και ένα άλλο σημείο που σχετίζεται με την εποπτεία. Όπως σας είπα, η διευκόλυνση ε, εισαγωγής αυτών των ειδών θα έχει ως αντίκτυμο την εποπτεία των εγκαταστάσεων έτσι ώστε να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές όπως ορίζουν οι εμπειρογνώμονες. Υπ' αυτή την έννοια προτείνεται μία νέα παράγραφος όπου αναφέρεται τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την επαλήθευση και εποπτεία της συμμόρφωσης των ε, κλειστών εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας με τις προδιαγραφές όπως ορίζονται από τον ορισμό της κλειστής εγκατάστασης έτσι ώστε και οι ενδεχόμενες μεταφορές να γίνονται κατά τρόπο έτσι ώστε να μην υπάρχει ε, απώλεια ξενικών ειδών και ειδών που δεν είναι στοχοθετημένα. Πρόκειται για τροπολογίες που είναι πολύ περιορισμένες. Νομίζω ότι θα πρέπει να τύχουν συνένεσης και το Συμβούλιο και η Κομισιόν συμφώνησαν και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία από την νομική υπηρεσία, τη γραμματεία το Συμβούλιο καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντάλλαξα απόψεις με ορισμένους σκιώδεις και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για να προωθήσουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και να βελτιώσουμε την πρόταση η οποία σας έχει υποβληθεί. Ευχαριστώ. Okay, thank you very Ευχαριστώ. Ε, για την έκθεση τον κύριο Φερέρα. Έχω δύο άτομα που μου ζητούν το λόγο. Ο κύριος Αρσένης πρώτος. Thank you very Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα διότι ε, έχουμε διάφορα είδη τα οποία απειλούνται από τους κανόνες της βιοπικιλότητος και ε, θεωρώ ότι η έκθεση του κυρίου Φερέρα είναι πολύ καλή, ε, βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε δύο θέματα τα οποία εντόπισε ο κύριος Φερέρα. Καταρχήν να υπάρχει ένα κλειστό σύστημα το οποίο να είναι επίγειο, ε, επί και επίσης να υπάρχει μία σοβαρή παρακολούθηση όλων αυτών των κλειστών συστημάτων κατά τρόπον ώστε να μπορέσει να υπάρξει σεβασμός των κανόνων. Συμφωνώ καταρχήν με όλες τις τροπολογίες οι οποίες υποβληθήκανε και που θα συζητηθούν στην πολιτική μας ομάδα για να δούμε εάν θέλουμε να περιλάβουμε ε, άλλες τροπολογίες. Καταρχήν όμως συμφωνώ με την έκθεση όπως παρουσιάστηκε. Ευχαριστώ. Ένα σύστημα κλειστό πρέπει υποχρεωτικά να είναι ε, στην ξηρά διότι η Ισπανία μας είχε προτείνει να ε, ε, κατασκευάσει ένα πλοίο το οποίο θα μπορούσε ε, να έχει χώρο να προετοιμάσει τα ψάρια και ε, μετά να τα τοποθετεί εις ε, τη θάλασσα όπου υπήρχαν ε, ισχυρά ρεύματα. Οπότε δεν είναι υποχρεωτικά αναγκαίο να είναι επί της ξηράς το σύστημα. Δεν, είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω αρκετά καλά, αλλά από ό,τι, ό,τι προσπάθησα να διερευνήσω ε, στην Ελλάδα όλοι μου είπαν ότι είναι ο πιο ασφαλής ε, τρόπος, δηλαδή να υπάρχουν ε, συστήματα στην ξηρά. Παρόλο που αντιλαμβάνουμε ότι έχουμε σπάνια ατυχήματα, αλλά εάν το πλοίο είχε κάποιο ατύχημα τότε δεν θα ήταν τόσο ασφαλές το σύστημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Διότι η πρόταση αυτή της Επιτροπής είναι μία πρόταση για την οποία μιλούμε για πολύ περισσότερα από τον ορισμό της κλειστής εγκατάστασης ιδιοκοτέρης. Κυρίως μιλούμε για λιγότερη γραφειοκρατία. Και αυτό είναι καλό. Πάντα είναι καλό κάτι τέτοιο, διότι σημαίνει λιγότερες προστάθειες για αυτούς που χρειάζονται τα συστήματα και μικρότερη οικονομική θυσία. Τώρα, εκτός από το νομικό πλαίσιο το οποίο θα εφαρμοστεί, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε Αν δεν κλείσει, δεν μπορώ να μιλήσω. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι κυρίως να αυξήσουμε την ασφάλεια και θα πρέπει να προσέξουμε ώστε η ενίσχυση της ασφάλειας να μην σημαίνει ότι θα πρέπει να αναλάβουμε άλλες δραστηριότητες που δύσκολα θα φέρουμε σε πέρας. Θα πρέπει λοιπόν την ασφάλεια να εξασφαλίσουμε χωρίς υπερβολικό συμπληρωματικό κόστο. Τώρα θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για μια αποχρώσα διαφορά. Κάποια στιγμή γίνεται λόγος για εγκαταστάσει ιχθυοκαλλιέργειας, καλύτερα να μιλούμε για το υδατοκαλλιέργεια, που είναι πιο ευρεία ω έννοια από την ηχθειοκαλλιέργεια, διότι μπορούμε να... Όταν μιλάμε για υδατοκαλλιέργεια περιλαμβάνουμε και τα άλλα θαλάσσια είδη, τα μαλάκια κτλ. Ούτως ή άλλως κατά τα άλλα συμφωνούμε με την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. η κυρία Μεντίνα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φερέιρο για την έκθεσή του, για την πρόταση αυτή της Επιτροπής. Οι, Επιτροπέ, οι υπηρεσίες της Επιτροπής λαμβάνουν υπόψη όλες τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, τις μελετάμε και κυρίως της τροπολογίας για την ε, προσαρμογή της νομικής βάσης και την χρησιμοποίηση για τις νέες συνθήκες που ισχύουν μετά θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνης σε διάφορα άρθρα. Τα λαμβάνουμε υπόψη, δεν μπορούμε να αποφανθούμε για αυτά τα θέματα ακόμη, δεδομένου το θέμα είναι ευαίσθητο, το μελετάμε, το σκεφτόμαστε ακόμη Τώρα, όσον αφορά άλλες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Σε πρώτη ανάλυση, έχουμε την εντύπωση ότι κάποιες από αυτές οι οποίες συζητήθηκαν και σε επίπεδο Συμβουλίου στρέφονται προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορούν να βελτιώσουν το κείμενο της Επιτροπής. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην τροπολογία που λέγει ότι θα πρέπει σε προθεσμία έξι μηνών να δημοσιεύει το κατάλογο των κλειστών εγκαταστάσεων. Τώρα, όσον αφορά για τις χερσαίες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, καταρχήν μας φαίνεται ότι αυτό ήταν προφανές. Άρα θα πρέπει να το αναλύσουμε πιο λεπτομεριακά, αλλά όπως σας είπα, καταρχήν Σωστά είναι τα πράγματα. Όσον αφορά την τροπολογία 5, στην οποία γίνονται κάποιες αλλαγές της ορολογίας για να μιλήσουμε για απώλειες βιολογικού υλικού και ατόμων όπως λέγεται ή άλλων οργανισμών ε, συμφωνούμε Δεδομένου ότι εδώ καταρχάς εμείς είχαμε προβλέψει κάποιες βιολογικές κυρίως απολύσεις. Τώρα, το να συγκεκριμενοποιήσουμε σε περίπτωση πλημμύρας και τα αριθμό των μιλίων των χιλιόμετρων, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμο, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στον ορισμό, δεδομένου ότι ο ορισμός θα πρέπει να είναι γενικός και να μην κάνουμε εξειδίκευση όλων των μέτρων που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να μειώσουμε, να παρεμποδίσουμε τις απώλειες του βιολογικού υλικού των άλλων οργανισμών, έτσι όπως αναφέρονται στον ορισμό. Όσον αφορά την τροπολογία 6 για τον έλεγχο, θεωρούμε και την εποπτεία ότι τα κράτη-μέλη όντως είναι υπεύθυνα για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των άνθρων του κανονισμού αλλά μου φαίνεται ότι είναι κάπως επαναληπτική αυτή η τροπολογία αυτών που λέγονται στο άρθρο 1 του κανονισμού. Θα πρέπει να κάνουμε επαλήθευση αν από νομικής πλευράς είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η επανάληψη. Προς το παρόν αυτές τις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ. Και θα ήθελα τώρα να ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Φερέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αρχίζοντας θα ήθελα να χαιρετήσω την ε, παρουσία συνεδρίασή μας μιας ομάδας επισκεπτών αλλιέων από την Πορτογαλία που επισκέφτονται σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ήρθαν σήμερα στη συνάντηση της Επιτροπής μας. Πολλοί από αυτούς γνωρίζω ότι παρακολουθούν εκ του σύνεγγες και με μεγάλη προσοχή τις συζητήσεις που κάνουμε και κυρίως ε, τη θέματα που αφορούν τη μεταρρύθμιση κοινή αλληλευτικής πολιτικής και θα ήθελα να τους ε, χαιρετήσω και πάλι να τους καλωσορίσω και να τους ευχηθώ ευχάριστη και χρήσιμη διαμονή στι Βρυξέλλε και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, όσον αφορά τα σχόλια τα οποία έκαναν οι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου τον Ισκιάδη γιατί καθώς και την Κομισιά για τα σχολιά της σε σχέση με τις παρατηρήσεις πιστεύω ότι υπάρχουν ε, κοινέ θέσεις όσον αφορά τους στόχους του κοινωνικού. Τι θέλουμε να κάνουμε. Να εξασφαλίσουμε ε, μείωση της ε, μη απαραίτητης γραφειοκρατίας και του άχθους για όλους όσους απασχολούνται στον κλάδο αυτό. Δεύτερον, βλέπω ότι όλοι συμμερίζονται αυτή την γενική αρχή. Από εκεί και μετά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κάποια επιμέρους ε, θέματα στα οποία έχουμε διαφορές για να μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε σε κοινά λύσεις αποδεκτές από όλους. Διευκόλυνση δηλαδή του γραφειοκρατικού άχθους και της αρχής της εισαγωγής καθώς και διασφάλισης του περιβάλλοντος. Όσον αφορά κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν σε σχέση με το αν είναι υποχρεωτικό τα κράτη-μέλη να κάνουν εποπτεία και έλεγχο των εγκαταστάσεων, των κλειστών για να δουν εάν συνάδουν με τις, τα προαπαιτούμενα δεν θεωρώ ότι είναι σε επανάληψη αυτό, δεδομένου ότι θέλουμε κυρίως να ευαισθητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη, να διασφαλίσουν το περιβάλλον, τις προβλήματα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν. Άρα δεν το θεωρώ ως επανάληψη, αλλά ως διευκρίνηση. Και νομίζω ότι αυτό αιτιολογείται, δεδομένου ότι κάνουμε εδώ τον ορισμό της κλειστής εγκατάστασης δίδατο κάνουμε την εισαγωγή αυτών των ξενικών ειδών. Εν πάση περιπτώσει, εάν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε και περαιτέρω. νομίζω ότι είναι ε, χρήσιμο να υπογραμμιστεί και πάλι αυτή η υποχρέωση των κρατών Τώρα, αφορά το δικό σας σχόλιο, σαν αφορά την ε, ύπαρξη άλλων εγκαταστάσεων και όχι μόνο χερσαίων, θα πρέπει να δούμε σύμφωνα με τις επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις τι προβλέπετε η τροπολογία αυτή όμως έχει ειδικά να κάνει με τις χερσαίες κλειστές εγκαταστάσεις δατοκαλλιέρωσης, όπως είπε και προηγουμένως η εκπρόσωπος της Κομισιόν. Η τροπολογία, την νομοθετική, γίνεται λόγος για τον ορισμό αυτών των εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη την, ε, το ίμπας. Εδώ ε, για αυτές μιλούμε σύμφωνα με το ΙΜΠΑΣ. Και ξέρουμε ότι, όπως σας είπα, με την υποστήριξη των τεχνικών και επιστημονικών εξελίξεων θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες μετατροπές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Φερέιρα. Ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τους επισκέπτες μας από την Πορτογαλία που είναι ένα από τα πολύ σημαντικά κράτη για την αλία της Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε. Πρέπει να σας πω ότι έχετε Πορτογάλους ευρωβουλευτές που παρακολουθούν ιδιαίτερα και ενδιαφέρονται για το θέμα της αλίας. Λοιπόν, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για την έκθεση Φεραίρα 7 Μαΐου, Παρασκευή. Έγκριση του σχεδίου έκθεσης στη συνεδρίαση της Δευτέρας Ιουνίου και συζήτηση και ψηφοφορία στην ε, Ολομέλεια ή στις, ε, τον Ιούλιο του Σεπτέμβριο. Επόμενο σημείο της Σχέδιο προπολογισμού του 2011. Τμήμα 3. Επιτροπή. δεν προβλέπονται σε επίπεδο Επιτροπή Πολιτική Αλλαγή σύμφωνα με τη Συνθήκη Λισαβόνα. Έχει εγκρίνει τον Απρίλιο τον προπολογισμό και όχι το σχέδιο προπολογισμού όπω στο παρελθόν. Το Συμβούλιο θα μα εξηγήσει την ε, θέση του στι 15-16 Ιουλίου. Η Επιτροπή Αλληλεία θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για το σχέδιο προπολογισμού 2011 και να καταθέσει. Now, this... Η έκθεση αυτή γνωμοδότησης έχει ανατεθεί στην κυρία Ρόντοστ. Και το χρονοδιάγραμμα δύσκολα πάντα ε, γίνεται δεδομένου ότι έχουν τις καλοκαιρινές διακοπές αλλά εν πάση περιπτώσει η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 21 21η Ιουλίου Επιτροπή ε, Αλίας, ψηφοφορία 30 Αυγούστου, εκ μέρους της ε, Επιτροπής, ο κύριος Τζόνσον θα μας παρουσιάσει την απόφαση της Επιτροπής μετά από την έγκρισή του από το σύνολο των ε, Επιτρόπων την 27η Απριλίου και μετά την παρουσίαση που θα γίνει από τον κύριο Τζόνσον θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρόντος και σε άλλους συναδέλφους που θέλουν να λάβουν το λόγο. Κύριε Τζόνσον από την Μάρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προτού ξεκινήσω να παρουσιάσω την λεπτομερή πρόταση που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της αλληλείας και των ναυτιλιακών υποθέσεων, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα βασικά σημεία, διότι βρισκόμαστε φέτος σε μία νέα δημοσιονομική διαδικασία και είναι η πρώτη φορά που ο προϋπολογισμός θα υιοθετηθεί βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας και υπάρχουν υπάρχουν ε, διαφορές με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαμε στο παρελθόν. Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει εισάγει μία καινοτομία η οποία θα επιταχύνει τη διαδικασία διότι θα υπάρχει φέτο μόνο μία ανάγνωση ενώ στο παρελθόν είχαμε ε, δύο αναγνώσεις στο Κοινοβούλιο και δύο ε, στο Συμβούλιο. Και ένα άλλο πολύ βασικό θέμα είναι ότι ε, θα είναι ισότιμο το Συμβούλιο για το Κοινοβούλιο στα θέματα του προπολογισμού. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή πλέον υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές ε, δαπάνες όπου το Συμβούλιο θα είχε τον τελευταίο λόγο σχετικά με τις υποχρεωτικές δαπάνες και το Κοινοβούλιο στις μη υποχρεωτικές αλλά οι δύο δημοσιονομικές αρχές θα χρειαστεί να συμφωνήσουν Αφού λοιπόν υπάρξει μια ανάγνωση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, εάν υπάρχει μια διαφορά θα υπάρξει μια Επιτροπή Συνδιαλλαγής η οποία θα έχει τρεις εβδομάδες για να συμφωνήσει. Ελπίζουμε στο τέλος των τριών εβδομάδων με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Οπότε, εάν όμως αυτό δεν επιτευχθεί, θα χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώσει νέες προτάσεις. Όπως σας είπα την περασμένη εβδομάδα, 28 Απριλίου, υιοθετήσαμε το σχέδιο προϋπολογισμού και παρουσίασε ο κύριος Λεβαντόφσκι το θέμα στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και νομίζω ότι η Επιτροπή Ελίες είναι η επόμενη επιτροπή η οποία ενημερώμενε σχετικά με το νέο προϋπολογισμό. Θα ήθελα να αναφερθώ γενικά στον προϋπολογισμό προτού επισέλθω σε λεπτομέρειες. Προτείνουμε 142,6 δις ε, όσον αφορά τις ε, ε, δεσμεύσεις και εξ αυτών έχουμε 130 εκατομμύρια τα οποία αντιπροσωπεύουν ε, όσον αφορά τις πληρωμές 130 εκατομμύρια που αντιπροσωπεύουν αύξηση σε σχέση με το παρελθόν. Βεβαίως για όσους δεν είναι έμπειροι στο θέμα δεν είναι προφανείς οι διαφορές διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να δεσμευθεί νομικά να ε, χρηματοδοτήσει υπό προϋποθέσεις. Ε, όσον αφορά τις δεσμεύσεις ε, ε, και τη διαφορά τους από τις πληρωμές είναι ότι το δεύτερο αναφέρεται σε καταβολές που θα γίνουν στο τρέχον έτος. Οι δεσμεύσεις όμως χρειάζονται για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να ε, μεταφέρουν χρήματα προς τις Βρυξέλλες για να μπορέσουν να ε, γίνουν σεβαστές οι δεσμεύσεις που έχουν αναλυθεί. Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ελπίζουμε κατά τον Οκτώβριο. Όσον αφορά την ε, αλληλεία και την ναυτιλία ο προϋπολογισμός είναι πιο περιορισμένος. Προβλέπουμε να υπάρχει μία συνέχεια δράσεων και προγραμμάτων ε, υπάρχει βασικά σταθερότης και τα ποσά για το 2011 είναι ευθυγραμμισμένα με ε, το, τα ποσά που υπήρχαν στον προϋπολογισμό του 2010. Σύνολο ε, προς, προβλέπουμε σε ε, δεσμεύσει 996,5 εκατομμύρια και αν θέλετε να δείτε όλες τις προτάσεις θα δείτε ότι αυτό αντιπροσωπεύει 7% του προϋπολογισμού του συνολικού ε, ενώ οι ε, πληρωμές έχουν μία αύξηση 6,3% και όπως σας είπα αυτά τα ποσά συνάδουν με αυτά τα οποία υπήρχαν στον προϋπολογισμό του 2010. Όπως σας είπα είναι πολύ βασικό να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει μία καλή βάση στις προτάσεις μας και γι' αυτό ε, ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένοι υπολογισμοί σχετικά με τις δεσμεύσεις που θα αναλυφθούν ε, φέτος και ε, θα εμποδίσουμε στο τέλος του έτους να υπάρχει ε, ανεπαρκής εφαρμογή του προϋπολογισμού που θα ήταν κρίμα ιδίω σε ε, δύσκολες ημέρες σαν δηλαδή το να μεταφέρουν τα κράτη κεφάλαια που δεν θα χρησιμοποιηθούν σε αυτές τις δύσκολες ημέρες δεν θα ήταν καλό. Το πιο ο, βασικό, ο, πιο βασικός τομέας δαπανών είναι στην, ε, ε, ε, την αλληλεία στο κεφάλαιο 11.6 όπου το Ταμείο Αλληλείας αντιπροσωπεύει δύο τρίτα της Γενικής Διευθύνσεως ΜΑΡΕ. Δηλαδή το 2011 προτείνουμε μία αύξηση 2% σε 657 εκατομμύρια από 643 εκατομμύρια που ήταν το 2010. Βεβαίως δεν ε, έχουμε ευχέρεια στο ποσό το οποίο προσφέρουμε διότι πρόκειται για ένα διαρθρωτικό ταμείο και το ποσό το οποίο ε, ε, διατίθεται από το 2007 στο 2013 είχε αποφασιστεί στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005. Επιπλέον βέβαια τα κράτη-μέλη έχουν ε, καταρτήσει τα προγράμματά τους γνωρίζοντας τι ποσά προτείνονται και αυτά τα λειτουργικά προγράμματα έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχει ε, ε, μία συνολική ε, αποδοχή του επταετούς προγράμματος και άρα υπάρχει δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επταετία η οποία πρέπει να πληρώνει τις ετήσιες δόσεις των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η ευθύνη για την καθημερινή εφαρμογή του προγράμματος έχει αναλυθεί από τα κράτη τα οποία θα επιλέξουν τους αποδέκτες, θα καθορίσουν τις δράσεις και είναι υπεύθυνα για την καταβολή των ποσών κατευθείαν εις τους αποδέκτες θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στο Ταμείο Αλίας έχουμε τα 567 εκατομμύρια που ανέφερα και θα καλύψουν όλες τις δράσεις. Ε, ε, έχουμε 463 εκατομμύρια τα οποία θα διατεθούν διότι το Λουξεμβούργο ε, δεν έχει πρόγραμμα για, στα πλαίσια του Ταμείου Αλληλείας και επιπλέον υπάρχει και ένα ποσό για να κλείσει η προηγούμενη ε, περίοδος προγραμματισμού δηλαδή η περίοδος 2002-2007 η οποία κλείνει τώρα δηλαδή ορισμένα τελικά έγγραφα έχουν ληφθεί ήδη από ορισμένα κράτη-μέλη και μέχρι το Σεπτέμβριο ελπίζουμε ότι θα έχουμε ολοκληρώσει το φάκελο και έτσι θα μπορέσει να προχωρήσει η ρευστοποίηση και το κλείσιμο το πιο βασικό θέμα είναι το θέμα της διεθνούς αλίας και υπερποντίου ε, ε, αλίες που εκπροσωπεί το 16% του προπολογισμού που έχουμε προϋπολογίσει για το 2011 και καλύπτει τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες ε, ε, αλληλείας και ε, την στήριξη του τομέα που υπάρχει σε όλες τις συμφωνίες για το 2011 θα πληρώσουμε για τις συμφωνίες που θα εφαρμοστούν το 2011 αλλά και επίσης και για τις συμφωνίες οι οποίες θα τύχουν αναδιαπραγμάτευση το 2011 και αυτές θα καλυφθούν από το ποσό του 2011. Τα θέματα αυτά δεν εμφανίζονται στη γραμμή του προϋπολογισμού αλλά σε ένα αποθεματικό ε, του προϋπολογισμού ε, έχουμε προτείνει 165 ε, εκατομμύρια που είναι μία μείωση από τα 174 εκατομμύρια που έχουμε φέτος και όσον αφορά τις ε, πληρωμές ε, έχουμε 159 εκατομμύρια που είναι και πάλι μία μείωση έναντι των 172 εκατομμυρίων που υπάρχουν για εφέτος. Ε, ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει μία μείωση εις ε, τις ευκαιρίες αλληλείας σύμφωνα με τις συμφωνίες και ελπίζουμε το 2011 να έχουμε ε, ίδιες, ίδιο αριθμό συμφωνιών σαν αυτές που ισχύουν για το 2010. Το επόμενο πιο βασικό θέμα είναι ο έλεγχος και εδώ έχουμε προτείνει ένα ποσό 56,6 εκατομμυρίων ευρώ ε, ενώ το 10 είχαμε 53 κρόμητρια ε, ε, πράγμα το οποίο σημαίνει μία αύξηση 5,5% και στις πληρωμές έχουμε μία σημαντική αύξηση από 40 σε 46 εκατομμύρια το 2011. Ο, το κεφάλαιο αυτό το 1108 προβλέπει δύο είδη δαπανών αρχικώς τα προγράμματα προγράμματα ελέγχου που θα εφαρμοστούν στα κράτη-μέλη όπου δηλαδή τα κράτη-μέλη θα αναλάβουν την ευθύνη για τον έλεγχο και την εφαρμογή της πολιτικής αλληλείας, άρα τα κράτη-μέλη θα προβούν εις τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις και θα χρειαστεί να επανδρωθούν με τα αναγκαία μέση ε, για να προβούν εις τις επιθεωρήσεις και θα συγχρηματοδοτήσουμε ορισμένα από αυτά τα μέσα. Υπάρχει και ο κανονισμός ελέγχου που ισχύει πλέον, που αναφέρεται στις νέες κατηγορίες πλοίων και ενθαρρύνει επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και η μικρή αύξηση σε αυτή τη γραμμή του προϋπολογισμού αποβλέπει ε, την ρύθμιση αυτού του επιπλέον, ε, ε, αυτής της επιπλέον δαπάνης. Επίσης υπάρχει και το γραφείο ελέγχου στο Βίγκο και όπως όλοι οι οργανισμοί που έχουν καταρτιστεί σε ε, κοινοτικό επίπεδο συμβάλλει ή στην λειτουργία του οργανισμού αυτού ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και επειδή ε, ο οργανισμός αυτός ισχύει εδώ και δύο χρόνια βρίσκεται πλέον ε, σε ταχύτητα ομαλής πορείας έχει ε, καλυφθεί πλήρης πάντρωση υπήρχε τον προηγούμενο ο χρόνο ένα πλεόνασμα του προπολογισμού το οποίο όμως καλύφθηκε στη συνέχεια και ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μία μειωμένη μόνο αύξηση των ε, δαπανών που προβλέπεται της τάξης του 5% η διατήρηση το κεφάλαιο 1107 που καλύπτει ουσιαστικώς τα προγράμματα συλλογή στοιχείων, δηλαδή όπως κάνουμε για τον έλεγχο και την εφαρμογή στα κράτη-μέλη, θέλουμε ε, να καλύψουμε τα έξοδα που κάνουν τα κράτη για να ε, παρακολουθούν την πολιτική αλληλείας. Προβλέπουμε στο τομέα αυτό 50,5 ε, εκατομμύρια, μία ελάχιστη αύξηση αύξηση σε σχέση με το φετινό ποσό των 49 εκατονομία. Ζητάμε ε, όμως 45 εκατομμύρια για τις πληρωμές σε σχέση με τις 39 που είχαμε το 2010 και ε, όσον αφορά τα δύο τελευταία κεφάλαια τα οποία ανέφερα πρέπει να σας πω ότι θα υπάρχει μια καλύτερη χρήση των ε, κεφαλαίων επιτόπου, δηλαδή σε τομείς όπου είχαμε προβλήματα ή στο παρελθόν όσον αφορά την αφομοίωση και την εφαρμογή, έχουν ε, ληφθεί μέτρα για να τα αντιμετωπίσουμε και τώρα αποδίδουν και ε, αυτό εξηγεί γιατί ζητούμε να αυξηθούν ε, οι δεσμεύσεις μας στο τομέα αυτό. Μετά, όσον αφορά ε, το κεφάλαιο 1102 που είναι οι αγορές αλληλείες όπου υπάρχει η κοινή οργάνωση αγοράς για τα αλληλευτικά προϊόντα όπου καλύπτονται έξι συνολικά μέτρα και το άλλα μέτρα τα οποία υπάρχουν είναι η στήριξη των χρηστών εις τις απόμακρες περιοχές στην Πορτογαλία, στη Γαλλία και στην Ισπανία και ε, οι ε, δεσμεύσεις για τον ε, τομέα αυτό παραμένουν σταθερές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι όσον αφορά τις απόμακρες περιοχές το ποσό που προτείνεται κάθε χρόνια βασίζεται στη νομική βάση. νομική βάση και έχει καταρτήσει ένα σύστημα το οποίο προβλέπει ένα σύστημα κάπως χαμηλότερο από 15 εκατομμύρια που θα κατανεμηθεί στα τρία κράτη και τα οποία μπορούμε να προτείνουμε και είναι το μόνο το οποίο μπορεί να εκτελέσει σαν δέσμευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσο αναφορά τις περαιτέρω δεσμεύσεις έχουμε μία μείωση ε, σε σχέση με το 2010 και ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε αυτή τη μείωση είναι διότι εξετάσαμε την ιστορική εκτέλεση και όπως σας είπα σε αυτή την εποχή δεν θέλουμε να ζητήσουμε πόρους τους οποίους δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε. Τέλος όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Το κεφάλαιο της διακυβέρνησης είναι μικρό αλλά σημαντικό διότι σύμφωνα με το κεφάλαιο αυτό καλύπτουμε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται το διάλογο με τους ενδιαφερομένους ε, από την κοινή αλληλευτική πολιτική και ε, προβλέπουμε και χορηγήσεις οι οποίες επιτρέπουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, προετοιμάζεται και να συμμετέχει στην ΑΚΦΑ. Ε, το ποσό είναι 6,4 ε, εκατομμύρια στις δεσμεύσεις και 5,8 εκατομμύρια εις τις πληρωμές και τέλος θα μιλήσω για την αυτιλιακή πολιτική. Η μόνη σχέση που έχουμε αυτή, με αυτό το θέμα τώρα είναι οι δεσμεύσεις πληρωμών διότι 8, 9 και 10 είχαμε είχαμε καταρτήσει πιλωτικές ενέργειες τις οποίες εκτελούσαμε και είχαν περιοριστεί σε δύο έως τρία χρόνια. Άρα αυτή τη στιγμή δεν ζητούμε νέες δεσμεύσεις διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νομική βάση. Αυτό το οποίο ζητούμε είναι 5,4 εκατομμύρια σε δεσμεύσεις πληρωμών για να συνεχιστούν οι δράσεις οι οποίες εκτελούνται και καταρτίζουν με μια νέα νομική βάση για την ναυτιλιακή πολιτική η οποία ε, είναι αρκετά προχωρημένη αλλά μέχρι ότου ολοκληρωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν μπορεί να κάνει πρόταση πρέπει πρώτα να ε, έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν είμαστε σε θέση να καλυφθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τζόνσον για την σαφέστατη αυτή παρουσίαση uh, και χαίρομαι ε, για τη διεξοδική παρουσίαση. Τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Ρόνταστ. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, αλλά ιδιαίτερο τον κύριο Τζόνσον. Ξέρω ότι η παρουσίαση ενός προϋπολογισμού είναι πάντοτε μία οδυνηρή ε, υπόθεση αλλά παρουσιάσατε σωστά το θέμα ε, και ε, παρόλα αυτά θα ήθελα να σας κάνω ορισμένες ερωτήσεις και ελπίζω θα μπορέσετε να μου απαντήσετε. Η πρώτη μου ερώτηση είναι δύο ουσιαστικές ερωτήσεις. Δηλαδή, είπατε στην ομιλία σας δεν είπατε μάλλον τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τουλάχιστον εγώ δεν κατάλαβα ποιες είναι οι προτεραιότητες σύμφωνα με την παρουσίασή σας διότι εσείς πήγατε ε, από ε, τη σειρά των αριθμών και όχι τη σειρά των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή ε, πώς θα, αντικαταστρώ θα θα εμφανιστούν ή στο πρόγραμμα του 2011 οι προτεραιότητες αυτές. Επίσης όσον αφορά το ταμείο το οποίο περάσατε εντάχει θα ήθελα να ρωτήσω πόσο ακόμη θα υπάρχουν ε, πόροι με από το παλιό μέσο που χρησιμοποιήσουμε και μετά θα κάνω ερωτήσεις για το 11 0301 διεθνείς συμφωνίες όπου οι αριθμοί δεν είναι σαφείς ακόμη και αν συμπεριλάβει κανείς τα αποθέματα διότι σε αυτή την πολιτική παρουσίαση η Επιτροπή λέγει ότι θα υπάρξουν μειωμένες πληρωμές σας παρακαλώ ε, για ποιες ε, συμφωνίες μιλάτε και γιατί θα υπάρξουν μειωμένες πληρωμές μετά, όσον αφορά το 11.06.02 γιατί στο κεφάλαιο 11 υπάρχει μία γραμμή για την προώθηση της συμφιλιώσεως στη Βόρειο Ιρλανδία. Τι σχέση έχει αυτό με την πολιτική αλίας. Εγώ δεν το καταλαβαίνω Τρίτο ερώτημα, όσον αφορά το 11.702 ε, στήριξη των πόρων αλληλείας για την βελτίωση της, ε, ε, της εμπειρίας γιατί έχουν μειωθεί τα ποσά εδώ τα οποία δεν είναι βίωνο για μια ικανοποιητική πολιτική αλληλείας δεν θα υπάρξει δηλαδή καλή πολιτική αλληλείας υπό αυτές τις προϋποθέσεις και τώρα έρχομαι στο 110805 τον ε, οργανισμό ελέγχου που θα λάβει ένα εκατομμύριο περισσότερο το 2011 κάτι μας εξηγήσετε αλλά δεν το πολύ κατάλαβα μας είπατε δηλαδή ότι ε, υπήρχε ένα πλεόνασμα το 2009-2010 το οποίο δηλαδή στο 2010 καλύφθηκε αλλά το 2011 θα χρειαστούν και άλλα χρήματα θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς δημιουργήθηκε αυτό το ποσό και ε, σε τι θα χρησιμεύσει, πού θα εφαρμοστεί. Και τελευταίο ερώτημα όσον αφορά τον κανονισμό ελέγχου που αναφέρεται το σύστημα το ο σύστημα ελέγχου της ναυσιπλοείας τα πλοία πέραν των 15 μέτρων θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο είναι δαπανηρό και αντιλαμβάνομαι ότι η χώρα μου δεν έχει πλέον πόρους για να καλύψει τις ανάγκες του 2010. Τι θα γίνει, θα υπάρξουν επαρκείς πόροι για το 2011 σας ευχαριστώ και προσβλέπω σε μια θετική απάντηση. Ευχαριστούμε κυρία Ροντάστ. Ο κύριος Ζωμέρα ζήτησε το λόγο. Μία ερώτηση θα ήθελα, να υποβάλω σε σχέση με τον εποπτικό έλεγχο, το δίκτυο εποπτείες. Από όσο γνωρίζω και θα ήθελα να το επιβεβαιώσω, φαίνεται ότι επιτεύχθηκε μία, ε, ένα συμβιβασμός ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει ε, αυτό το δίκτυο, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Έχει γίνει ή όχι και αν όχι, γιατί δεν έγινε αυτή η χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φερέρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την διεξοδική παρουσίαση της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ. Νομίζω ότι πρόκειται, για μία έκθεση ύψης της σημασίας αυτή της κυρίας Ρόνταστ. Γιατί ό,τι συζητήσαμε σε αυτή την Επιτροπή έχει επιπτώσεις, επιπτώσεις δημοσιονομικές. Και υπ' αυτή την έννοια ο προϋπολογισμός είναι το μέσον που μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε πολλά από τα οποία συζητήσαμε. Χωρίς να προδικάσω ως προς τα αριθμητικά στοιχεία που μας δόθηκαν, γιατί θα εξεταστούν, καθώς και γενικά ζητήματα που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό καθεαυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν θα ήθελα να δώσω λεπτομέρειες. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για τα ανεπαρκή κονδύλια που έχουμε, για την ανεπαρκή χρηματοδότηση, αλλά αυτά είναι, αυτό είναι ένα γενικό σκεπτικό σε σχέση με το κεφάλαιο της αλίας. Απλώς θα ήθελα χωρίς να προδικάσω, να τονίσω αυτή την πτυχή και να εκφράσω την ανησυχία μας για την μείωση του προπολογισμού όπως προβλέπεται για την κοινή αγορά αλίες. Έχουμε κρίνει μεγάλες ανυπάρκειες και από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας είναι τα εισοδήματα των αλίων. Αυτό το συζητάμε κατ' εξακολούθηση. Από τότε που μιλήσαμε για τη μεταρρύθμιση της κοινή οργάνωσης αγορών της Αλίας. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, μπορέσουμε να παρέμβουμε ως προς τα έσοδα, το εισόδημα των αλλιέων και αυτό που βλέπουμε είναι μία μείωση για το επόμενο έτος είπε η Επιτροπή ότι υπάρχουν προβλήματα εκτέλεσης του προπολογισμού, αλλά αυτό μας δίνει ακόμα μεγαλύτερο δίκαιο ότι χρειάζεται μία μεταρρύθμιση της κοινή οργάνωσης αγοράς. Το να προσδίδεται σε αυτή την ε, αγορά λιγότερα κονδύλια ε, μας, ε, θα μας οδηγήσει σε επιδείνωση των προβλημάτων στο μέλλον. Αυτό ήθελα να πω ήδη από τώρα. Ευχαριστούμε κύριε Φερέ. Ο κύριος Γκάλαχερ. Καταρχήν να πω ότι η επεξήγηση του κύριου Τζόνσον ε, μπορεί να φαινόταν περίπλοκη, αλλά ήταν αρκετά απλή και για όποιον μπορούσε να καταγράψει τα στοιχεία. Μιλάμε για 7% ως προς τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Ο κύριος Τζόνσον δεν είναι εδώ να το αιτιολογήσει, απλώς μας αποστέλει αυτό το μήνυμα της απόφασης που ελήφθη από το Διευθυντήριο. Σε σχέση με τη θαλάσσια πολιτική 1109 μιλάμε για 7,4 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει νομική βάση, μας λέει. Αυτή η νομική βάση θα πρέπει να ισχύσει πριν γίνει η δέσμευση ή μπορούν να δαπανηθούν του χρόνου αυτά τα ποσά. Υπάρχει μια κάποια άλλη φόρμουλα για τη μεταβατική περίοδο. Μιλάμε για 56 εκατομμύρια ε, πιστώσεις υποχρεώσεων, αλλά είναι συγχρηματοδότηση. Τα 56 7 εκατομμύρια αφορούν συγχρηματοδότηση, δηλαδή και χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Και η ερώτηση είναι ίδια με το 1107 διατήρηση, όπου έχουμε μία αύξηση 14% σε 55 εκατομμύρια στις πληρωμές. Αυτό περιλαμβάνει και την χρηματοδότηση ε, από τα κράτη-μέλη, δηλαδή αφορά συγχρηματοδότηση. Ευχαριστούμε κύριε Κάλαχερ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω ορισμένα σχόλια. Φαίνεται από αυτά που μας λέτε κύριε Τζόνσον ότι ο συνολικός προϋπολογισμός θα αυξηθεί. Κατά 5% μας είπατε ή κάπως λιγότερο. Ενώ υπό τον τίτλο 11 βλέπουμε μείωση κατά 0,6% σε αυτούς τους καιρούς οικονομικής λιτότητας τον, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να υπάρξει αύξηση στις δαπάνες αλλά δεν θα ήθελα αυτοί που χάνουν να είναι οι αλληλείς να χάνουν από το διευθυντήριο. Μιλάτε για μείωση 20 εκατομμυρίων ευρώ ως προς τη χρηματοδότηση για συμφωνίες αλίας, δηλαδή για εταιρικέ συμφωνίες με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά μας είπατε ότι αυτό δεν σημαίνει λιγότερες δυνατότητες αλίευσης. Αυτό μου φαίνεται ένα θαύμα. Πώς ε, δαπανάτε 20 εκατομμύρια λιγότερα και να έχετε τα ίδια ποσοστά τα ίδια ποσά αλίας πέφτουν και οι τιμές βεβαίως των ειδών αλίας. Συμφωνώ με την κυρία Ροντάστ ότι τη στιγμή που οι ίδιοι αλεείς λένε ότι δεν υπάρχει επιστημονική έρευνα ούτε χρηματοδότηση, έτσι ώστε να έχουμε τις ε, πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να βασιστούμε ως προς την πληθώρα στοιχείων όπως τέλη, ποσοστώσεις, κιλοβάτ, κιλοβατόρες και ούτω καθεξής, το να μειώνουμε τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού ως προς τις επιστημονικές πληροφορίες είναι ο εντελώς λανθασμένος τρόπος. Άρα μας ανησυχούν ορισμένες πληροφορίες που μας δώσατε και βεβαίως η Επιτροπή θα έχει πολύ περισσότερα να πει κατά τη δημοσιονομική διαδικασία. Ίσως όμως μπορείτε να μας δώσετε ε, ορισμένες απαντήσεις. Σας δίνω το λόγο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στι περισσότερε ερωτήσει, έξω από κανένα δύο θέματα τα οποία δεν γνωρίζω πλέον και θα επανέλθουμε. Βεβαίω, θα ήθελα να τονίσω ευθύ εξ αρχή ότι πάντα μιλούμε για πρόταση τη Επιτροπή. Το Κοινοβούλιο είναι ένα από τα δύο κοινοτικά όργανα που έχει αρμοδιότητες και εξουσίες για τη λήψη απόφαση. Γι' αυτό πάντα υπάρχει περιθώριο. Αλλά θα ήθελα επίσης να ρωτήσω ότι όταν υποβάλλουμε μια πρόταση δεν την κάνουμε απομονωμένα αλλά στα πλαίσια ενός χρηματοδοτικού πλαισίου το οποίο καλυπτεί την περίοδο 2007-2013. Αυτό λοιπόν το δημοσιονομικό πλαίσιο έχει κεφάλαια και η αλληλεία και η ναυτιλία είναι στο κεφάλαιο φυσική πόρη. Εδώ έχουμε τις δαπάνες της γεωργίας, τις δαπάνες για το περιβάλλον, για την προσθήκη των κανετών, για την υγεία, καθώς και τις δαπάνες για τον τομέα της ναυτιλίας και την αλληλεία. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ε, διάφορα ποσά, τα οποία έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων αφορούν τα δύο τρίτα τα διαχρονικά μέρα για την αλληλεγγύη και διάρκεια όλες αυτής της ε, επταετίας έχουν κάνει διάφορα λειτουργικά προγράμματα τα κράτη-μέλη και τα εφαρμόζουν όπου χρειάζεται, αλλά αν υπάρχει κάποια εξέλιξη μπορεί να υπάρχουν και Τώρα, επανέρχομαι στην αρχική ερώτηση της ηγήτριας. Ποιες είναι οι προτεραιότητες της Επιτροπής, ρώτησε. Τις παρουσίασε συνολικά στα πλαίσια της παρουσίας του προορισμού του 2011 και βεβαίως υπάρχει προτεραιότητα στο δικό μας τομέα. Και όταν ο Επίτροπος ε, μίλησε στην Κόμπου την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι οι προτεραιότητες τις οποίες θέλουμε εμείς ε, να θέσουμε σε εφαρμογή είναι να ξαναρχίσουμε πάλι υποστήριξη αναθέρμανση της οικονομίας στην περίοδο μετά την κρίση για το 2011 και βεβαίως στρατηγική στόχη 2020. Και ξέρουμε ότι κάποια ποσά εντοπίστηκαν από την Επιτροπή για να συνεισφέρουν στην ε, ε, υλοποίηση των στόχων 2020. Τώρα, τι δική μας, το δικό μας το θέμα, το δικό μας κεφάλαιο, το δικό μας Οι προτεραιότητες αντικατοπτρίζονται στον τρόπο με τον οποίο σας έκανα την παρουσίαση. Σας παρουσίασα τις δαπάνες ανάλογα με την σημασία της σπουδαιότητα των διαφόρων κεφαλαίων. Και το πιο σημαντικό είναι για μας τα διαρθρωτικά μέτρα, εκεί που βλέπουμε να υπάρχει πολύ μικρή ε, αύξηση σε πλήρη συμφωνία με τα προγράμματα. Επίσης είδα ότι στο διεθνές κεφάλαιο, αν θέλετε, παρουσιάσαμε μικρή μείωση και είναι η στιγμή να παρουσιάσουμε το άλλο θέμα, όπως είπε και ο κ. Στίβενσον, γιατί προβλέπεται εδώ μείωση. Είναι σαφές ότι όταν κάνουμε διαπραγμάτευση εταιρικών συμφωνιών και θα κάνουμε πολλές με τρίτες χώρες, δεδομένου ότι έχουμε αυτή τη στιγμή πολλά ποσά τα οποία θα πάνε στο αποτελεσματικό του 2011 θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Ότι τα σχετικά πρωτόκολλα λήγουν ή κατά τη διάρκεια του παρόντος έτους ή θα ε, σταματήσουν να ισχύουν, θα λήξουν την αρχή της επόμενης χρονιάς, όποτε θα αρχίσει η διαπραγμάτευση για νέες συμφωνίες, νέα πρωτόκολλα. Είναι λοιπόν απόλυτα σαφές για μας ότι αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι ότι θα ξαναρχίσουμε διαπραγματεύσεις ακριβώς με στόχο να μην εξασφαλίσουμε ότι καλύτερο μπορούμε για τους πόρους που έχουμε, αλλά να κάνουμε σωστές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις τακτικής με τους εταίρους μας. Και οι προφορίες που έχω είναι ότι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε και αυτός είναι ο στόχος, τον ίδιο αριθμό εταιρικών συμφωνιών με τρίτες χώρες και τα πρωτόκολλα τα συνδέαμενα το 2011 με αυτά που έχουμε σήμερα και τις και να διατηρήσουμε τις δυνατότητες αλήψης τις ίδιες με φέτος. Βεβαίω το κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει απλώς και μόνο τις διεθνείς συμφωνίες αλίας, καλύπτει επίσης και μέτρα που έχουν σχέση με οργανώσεις διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο ή με θελούσιες συνεισφορές. Και υπάρχει μείωση διότι μία δράση η οποία έχει αναλυθεί διαχείριση σε περιφερειακό επίπεδο δεν θα συνεχιστεί το 2011. Και εδώ βεβαίω εξοικονομούμε περισσότερο 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, για να επανέλθω στι άλλε προτεραιότητε, τι υπόλοιπε. Έχουμε το θέμα τη θέση σε ισχύ και του ελέγχου που είναι κύρια προτεραιότητα και α είμαστε απόλυτα σαφεί για το τι κάνει ο δικό μα προπολογισμό. Στον έλεγχο της ε, στον τομέα του ελέγχου και την εποπτεία δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις δαπάνες ή ακόμη και μεγάλο μέρος των δαπανών που, που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη-μέλη για να φέρουν σε πέρα σε αυτή τη δραστηριότητα η οποία είναι τόσο πολύπλοκη και πολλές φορές αυτές οι δραστηριότητες είναι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν από κοινού πολλά Υπουργεία και, μόνο, και όχι μόνο το Υπουργείο Αλίας. Τι προσπαθούμε να κάνουμε εμείς με τα κονδύλια που διαθέτουμε. Να στοχεύσουμε τα σημαντικά θέματα στον τομέα αυτό και για μας αυτό που είναι σημαντικό είναι η αποδοτική εφαρμογή των ε, κανονισμών που αφορούν την εποπτεία και τον έλεγχο και προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την ε, ε, δημιουργία της τεχνολογίας που θα επιτρέψει στην εποπτεία να γίνεται αποτελεσματικά. Και εδώ φτάνω στο θέμα που έφυξε ο κύριος Κάλαγερ. τα ποσά τα οποία συμπεριλαμβάνονται εδώ. Συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά, τα ποσά χρηματοδότηση των κρατών μελών. Θα του πω όχι. Εδώ μιλούμε για αμυγός κοινοτικά κονδύλια ή στο 2008 ή στο 2007 και εδώ όταν μιλούμε για συλλογή δεδομένων, για τεχνική ενίσχυση ή για εποπτεία. Και εδώ σε αυτούς τους τομείς και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεισφέρουν με τις δαδικές κονδύλια έτσι όπως το ορίζει η νομοθεσία. Εδώ μιλάμε μόνο για κοινοτική χρηματοδότηση. Τώρα, επίσης, η συγγήτρια έθεσε ένα θέμα για την FIAFG και τη συνέχιση της. Κατά διάρκεια της παρουσίασή μου είπα ότι όντω για μας η FAFG βρίσκεται στην ε, τερματική της, στην τελική της φάση. Ξέρουμε ότι πρόκειται για κάτι το οποίο έχει τελειώσει η συμφωνία που έχει κυρωθεί από πέντε κράτη-μέλη. Έχουμε, θα πάρουμε τα σχετικά έγγραφα από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη το Σεπτέμβριο και το 2011 θα παραμείνει ένα μόνο Η μόνη πόροι μόνο εδώ θα είναι κονδύλια πληρωμής. Δεν θα δεσμευτούν άλλα κονδύλια για την FIFG. Και πρέπει να πω ότι οι πληρωμές πέρσι ήταν πολύ λιγότερες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, αυτό που είπατε και το θέμα της ε, συμφωνίας στην ίδια την δεν γνωρίζω καθόλου το θέμα αυτό, δεν πρέπει να το εξετάσω. Επίσης, εκφράσατε ανησυχίε για το θέμα της, ε, των επιστημονικών γνώσεων. Εμείς ε, συμμεριζόμαστε την άποψη ότι είναι θεμελιώδους σημασίες για να μπορέσει η όλη η στρατηγική στην αλληλεία να αποδοθεί σωστά. Και βλέπω του αριθμού όντω για τεχνική και επιστημονική βοήθεια όσον αφορά τις δεσμεύσεις από 5 εκατομμύρια πήγαμε στα 4,5 και όσον αφορά τις πληρωμές από 4,5 κατεβήκαμε στα 3,5 εκατομμύρια. Όπως εξήγησα και στην αρχή, οι πιστώσεις πληρωμών μας επιτρέπουν να κάνουμε τις διάφορες συμβάσεις και έχουμε μείωση 10% των κονδυλίων τα οποία μπορούμε να διαθέσουμε για τέτοιου είδους επιστημονική ε, σύμβουλη. Αυτό όμως είναι ένα μέλος μόνο της εικόνας. Αν δείτε την προηγούμενη γραμμή του προπολογισμού 11.07.01 που αφορά την συλλογή δεδομένων, θα δείτε ότι εδώ συγχρηματοδοτούμε τις δαπάνες των κρατών μελών όταν τα κράτη-μέλη συλλέγουν τα δεδομένα τα οποία χρημαζόμαστε για να εφαρμόσουμε την πολιτική μας. Και όντως όλοι το πλαίσιο συλλογή των δεδομένων πρέπει να πούμε ότι άλλαξε τα τελευταία δύο χρόνια και αυτό το οποίο έχουμε τώρα είναι ένα ε, πλαίσιο πιο αποδοτικό. Έχουμε τις επιστημονικές, ε, τα επιστημονικά δεδομένα που χρειαζόμαστε και αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε και αυτή ε, ήταν μία δική μας προτεραιότητα και επιλογή ή λοιπόν έπρεπε να συγχρηματοδοτήσουμε περισσότερο τα κράτη-μέλη που έκαναν αυτή τη δουλειά ή να κάνουμε διάφορες ε, συμβάσεις προμηθειών. Γι' αυτό εξηγείται αυτή η διαφορά. Πράγμα που δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε την απαραίτητη επιστημονική αρρωγή για να πάρουμε αποφάσεις. Τώρα, σε σχέση με τον οργανισμό, στο Βίγκο να φέρθηκε το πλεόνασμα του 2008 και είπαμε ότι στο 2009 μειώθηκε αυτό το πλεόνασμα σε σημαντικό βαθμό. Αν δείτε τις αριθμούς θα δείτε ότι έχουμε αύξηση του 5,5% στον προπολογισμό. Τι συνέβη το 2010 και στον προϋπολογισμό του 2010 τι είχαμε. Στο 8 και το 9 είχαμε σημαντικό πλεόνασμα τι έγινε με διάφορου διάφορους ότι το πλεόνασμα επανέρχεται στην διαδικασία του προπολογισμού. Ξαναμπαίνουν αυτά τα κονδύλια στο προπολογισμό. Και το 2010 το πλεόνασμα που δημιουργήθηκε το 9 και ξαναμπήκε στο προπολογισμό του 2010 ήταν 700 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λοιπόν μειώθηκε σημαντικά το πλεόνασμα και το ποσό που θα τεθεί πάλι και θα είναι φρέσκο χρήμα αν θέλετε στον προϋπολογισμό του 2011 είναι 185. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα φρέσκο χρήμα μισό και το μυρίου ευρώ το οποίο θα διατεθεί για την πλήρη λειτουργία του οργανισμού αυτού. Είδαμε λοιπόν να υπάρχει στον επιχειρησιακό της προϋπολογισμό και στον διοικητικό της προϋπολογισμό ε, εξελίξεις θετικές. Για ποιο λόγο, διότι τώρα έχει γίνει πλήρως ως αυτός ο οργανισμός στο Βίγκο. In to the, the actual increase... Σε σχέση τώρα με τις αυξομοιώσεις στον προπολογισμό, η σφαιρική αύξηση είναι 2,2 στον κοινοτικό προπολογισμό. Στον τομέα μας έχουμε περίπου σταθερά ποσά όσον αφορά δεσμεύσεις και πληρωμές. Έχουμε μια πάρα πολύ μικρή μείωση. Αν δούμε τους αριθμούς σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε ένα δις της δεσμεύσεις, φέτος έχουμε 1,96 και για τις κονδύλια πληρωμών, είχαμε τις πιστώσεις πληρωμών, είχαμε 800 και φέτος έχουμε 820 εκατομμύρια. Είμαστε λοιπόν σχεδόν σε κατάσταση σταθερότητας θα έλεγα. σε σχέση με την κοινή οργάνωση αγοράς. Κύριε Φερέα, σας επασχολεί η μείωση της χρηματοδότησης. Αυτό αφορά τις πιστώσεις πληρωμών. Δεν αφορά τις πιστώσεις δεσμεύσεων, οι οποίες είναι στο ίδιο επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Ότι εάν χρειαζόμαστε να κάνουμε πληρωμές πέραν των ποσών που διαθέτουμε στον προπολογισμό, θα βρούμε τρόπο να το κάνουμε. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Μέσω μεταφορών και μέσω άλλων μηχανισμών του προπολογισμού που έχουμε στη διαθεσή μας θα το κάνουμε. Όσον αφορά την διαθεσιμότητα του μηχανισμού να βοηθήσουμε τον τομέα, δεν θα υπάρξει αλλαγή μεταξύ των δύο αυτών. Και όσον αφορά τι απομακρυσμένε περιοχές, σας είπα ότι είμαστε σε ένα σύστημα όπου το ποσοστό βοήθειας που δίδεται στους παραγωγούς καθορίζεται από την νομική βάση και δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Ο κύριος Γκάλαχερ έθεσε το θέμα της συναχρηματοδότησης, το έθεσα το θέμα της ε, νομικής βάσης ε, επίσης για το 11.09. Τώρα, όσον αφορά τα 5 εκατομμύρια που προτείνει το 2011 είναι ότι έχουμε 5 εκατομμύρια για πιστώσεις πληρωμών και όχι για πιστώσεις δεσμεύσεων. Πρόκειται απλώς για πόρους οι οποίοι έχουν ε, σαφώς καθοριστεί για πληρωμές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δεσμεύει σύμφωνα με την, το νομικό πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα. Έχουμε κάποια ποσά για πιλωτικά σχέδια, αλλά όπως σας είπα, η διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργανείων είναι τριετής, γι' αυτό μέχρι να έχουμε μια νέα νομική βάση, ή όπως σας είπα, είναι κάτι το οποίο προχωρεί προπαρασκευαστικά στην Κομισιό, δεν θα μπορέσουμε να αναλάβουμε καμία νέα δράση. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να απαντήσω ερωτήσεις σας. Αν θέλετε σας ε, παράσχω περισσότερες προφορίες, κυρίως στο θέμα της ε, ε Βορειοϊρλανδίας. Και αν ε, μου ξέφυγε κάτι, ευχαρίστως να το συμπληρώσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τζόνσον για αυτή την πολύ σαφή παρουσίαση. Δεν ξέρω κατά πόσο κυρία Ρόνταστ θα ήθελε να έχει τον τελευταίο λόγο. Θα έχουμε συζητήσει και κατά τη διάρκεια του θέρους. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε κυρία Ρόνταστ. Όχι να προσθέσω. Ήθελα να ρωτήσω και πάλι τι γίνεται με το σύστημα ε, εποπτείας των οπλίων διότι δεν υπησύλθατε σε λεπτομέρειες, διότι τώρα είναι Μάιος εγώ είχα λάβει τις πληροφορίες τον Απρίλιο ότι δεν υπάρχει πλέον χρηματοδότηση για τον τομέα αυτό το οποίο χρειάζουμε εάν θέλουμε το 2014 όλα τα πλοία να έχουν εξοπλιστεί με αυτό το σύστημα παρακολουθήσεως. Τι θα γίνει αφού τώρα δεν έχουμε πλέον χρήματα, ισχύει αυτό, ε, θα υπάρχουν επαρκή πόροι για του χρόνου. Κύριε Τζόνσον, θέλετε να απαντήσετε παρακαλώ το θέμα με τον οποίο λειτουργεί η δαπάνη αυτή και ο έλεγχος ε, σημαίνει ότι ζητούμε να, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει τις προτεραιότητες θέσεις και σύμφωνα με τον νέο κανονισμό ελέγχου τα στοιχεία των δαπανών που συνδυάζονται με τις καινοτομίες που έχει καταρτήσει ο νέος κανονισμός ε, αποτελούν προτεραιότητες ε, προτεραιότητες. Ο τομέας για τον στον οποίο αναφέρεται δεν μου είναι γνωστός. Δεν έχουμε ακόμη υιοθετήσει τις πιστώσεις για το 2010 και φαντάζομαι ότι υπήρξαν άλλοι τομείς οι οποίοι θεωρήθηκαν ε, ότι ήταν μεγαλύτερης προτεραιότητας. Πάντοτε έχουμε περισσότερες αιτήσει από ό,τι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε και ο στόχος μας δεν είναι να τα χρηματοδοτήσουμε όλα, αλλά να είμαστε καταλήτης και να ενθαρρύνουμε τις ε, ε, δαπάνες ε, υπάρχει επίσης ε, ε, και ένα υψηλό ποσοστό συγχρηματοδοτήσεως. Όταν λοιπόν συγχρηματοδοτούμε με υψηλό συντελεστή συγχρηματοδότησης δεν διαθέτουμε τόσα χρήματα όσο υπό άλλες συνθήκες. Λοιπόν, 14 ε, και 15 Ιουλίου θα έχουμε μία συζήτηση για το σχέδιο της γνωμοδότησης. Οι τροπολογίες πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι τις 21 Ιουλίου και... Ε, υποθέτω ότι η ψηφοφορία θα είναι 30 Αυγούστου όταν θα γυρίσουμε δηλαδή από τις καλοκαιρινές διακοπές. Και Η συζήτηση επί του προπολογισμού θα γίνει 28 με 30 Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο έχουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι κυρία Ρόμπας και τώρα θα ήθελα να προχωρήσουμε στο θέμα 10, δηλαδή την ανταλλαγή με την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή πιλωτικών προγραμμάτων και προπαρασκευατικών δράσεων σε θέματα αλληλείας από το 2007 έχουμε καταρτήσει δύο προκαταρκτικές ε, ε, πολιτικές ε, όσον αφορά την ναυτιλιακή πολιτική και την προκαταρκτική την προκαταρκτική ε, ε, εκφώνηση και ε, μπορεί να υπάρξουν διάφορες μορφές δηλαδή οι δεσμεύσεις μπορούν να περιληφθούν στον προπολογισμό για τρία χρόνια και η νομοθετική διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από το τρίτο έτος. Υπήρξαν και δύο ακόμη ε, πιλωτικά προγράμματα για την αντικατάσταση των πλοίων για τον εμπορικό στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, υπάρχει ένα ε, περιγραμματικό πρόγραμμα για να εξετάσουμε την σκοπιμότητα και χρησιμότητα και μπορούν να υπάρξουν δεσμεύσεις για δύο συνεχή έτη και σήμερα η Γενική Διεύθυνση Αλίας θα αναφερθεί σε δύο γνώσεις, τέτοιες ενέργειες και θα δώσω τον λόγο στον κύριο Ρομπό της Γενικής Διευθύνσεως Αλίες. Ε, θαλάσσης, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε εδώ ίσως με κάποιες λεπτομέρειες γιατί είναι πρώτη φορά τη δράση αυτή η οποία αποβλέπει στην κατάρτιση μίας ε, ενός παρατηρητηρίου των αγορών της, ε, ε, των ε, προϊόντων της αλίας και της υδατοκαλλιέργειας. Σας είχαμε στείλει το Φεβρουάριο ήδη μία ενημέρωση για το πού βρισκόταν το θέμα και τώρα θα προσπαθήσω ίσως να μακρηγορήσω κάπως αλλά με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την πρωτοβουλία. Γι' αυτό πρώτα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ποιες ήταν οι ημερομηνίες που μας οδήγησαν στο να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Το δεύτερο είναι να σας υπενθυμίσω ταχαίως τους στόχους ενός τέτοιου παρατηρητηρίου και στη συνέχεια τις δραστηριότητες οι οποίες προβλέπονται στα πλαίσια αυτής της δράσης. Και τέλος, να αναφερθώ στο μέχρι που έχουν προχωρήσει οι εργασίες μας και να δώσω ορισμένες διευκρινήσεις για τις επόμενες φάσεις, για τους επόμενους μήνες και τα επόμενα έτη. Θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ σε ορισμένες βασικές ε, ημερομηνίες. Το καλοκαίρι του 2008 όπου η κρίση των καυσίμων και τα οικονομικά προβλήματα του τομέα της αλληλείας οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει μία ενημέρωση, μία ανακοίνωση στην οποία συμμετείχαν και το Κοινοβούλιο και ε, το Συμβούλιο και τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε την πρωτοβουλία να αποδώσει ένα προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ για να υπάρξει ένα παρατηρητήριο της αγοράς των προϊόντων αλληλείας και ε, υδατοκαλλιέργειας. Εκεί ανέρχεται αυτή η δράση και μόλις ελήφθη η απόφαση οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθύνθηκαν και στα κράτη-μέλη και στους κλασικούς συνεργάτες μας της βιομηχανίας ρωτώντας σας τι περιμέναν από αυτή τη γίνηση. Στείλαμε ένα ερωτηματολόγιο, αρχίσαμε ε, να αντιλαμβανόμαστε ε, τι ήθελαν οι διάφοροι οι διάφοροι ομολογοί μας από τους τομείς αυτούς. Οπότε από τον Ιούλιο του 2009 μπορέσαμε να εγγράψουμε το στόχο αυτό στο πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Σεπτέμβριο κάναμε έναν μειοδοτικό διαγωνισμό ο, ο οποίος τελικά κατεκυρώθη ένα γραφείο στο γραφείο ΚΟΖΕΑ για μία σύμβαση υπηρεσιών 3.935.000 ευρώ και μία διάρκεια 30 μηνών. Δηλαδή ε, σύμφωνα με τις συνθήκες που προαναφέρατε κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαστε στην αρχή αυτής της ε, δράσης και ίσως προτού προχωρήσουμε στις εργασίες ή στους επόμενους σταθμούς θα έπρεπε να σας υπενθυμίσουμε ποιοι είναι οι στόχοι αυτού του παρατηρητηρίου των αγορών των προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας. Σήμερα έχουμε το Eurostat, ένα οργανισμό ο οποίος μας δίνει ορισμένα εναρμονισμένα οικονομικά στοιχεία ευρωπαϊκά, αλλά και υπάρχει ένα αλλά, πρόκειται για ετήσια στοιχεία και παρουσιάζεται ένα μειονέκτημα. Δηλαδή, τα στοιχεία αυτά έρχονται πολύ ετεροχρονισμένα σε σχέση με την πραγματικότητα διότι ε, πρέπει καταρχήν να έχουν συγκεντρωθεί, να έχουν επαληθευθεί και διατίθενται ένα χρόνο μετά το συμβάν. Δεύτερον, η τα ε, στοιχεία της συγκυρίας, δηλαδή ε, καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία, τα οποία χρειάζονται που όπως σας είπα θα μας βοηθήσουν να παρακολουθήσουμε καλύτερα τον τομέα υπάρχουν αλλά είναι πολύ ετερογενή αναλόγως των χωρών. Αλλού υπάρχουν, αλλού δεν υπάρχουν και όπου υπάρχουν δεν είναι υποχρεωτικά συντονισμένα ή εναρμονισμένα. Άρα ο γενικός στόχος αυτού του παρατηρητηρίου είναι να διαθέσει στις ε, δημόσιες ε, αρχές και σε όλους τους ενδιαφερομένους του κλάδου ε, και στην εκπαίδευση και στην έρευνα, ε, πληροφόρηση οικονομική, τακτική και ε, σωστή όσον αφορά τις αγορές των προϊόντων αλληλείας και υδατοκαλλιέργειας και αυτό στο σύνολο της Ευρώπης και θα συνοδεύεται με τη δυνατότητα να υπάρξει σύγκριση της κατάστασης των διαφόρων αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και προς τα έξω και ε, πέραν αυτού εφόσον μιλάμε ε, για ε, οικονομική intelligence παρακολούθηση δηλαδή θα πρέπει να παρακολουθούμε όλες τις φάσεις από την πρώτη πώληση μέχρι την λιανοπόληση και βεβαίως και για τα εστιατόρια όπου χρειάζεται και να παρακολουθούμε τις κινήσεις των τιμών για τις εισαγωγές, εξαγωγές και μεταποίηση. Και ο τελικός στόχος αυτού του παρατηρητηρίου είναι να μπορέσει να ε, παρουσιάσει τη θέση της Ευρώπης από πλευράς προπτικής διεθνίους διότι όπως είπαμε και σήμερα το πρωί ε, όταν παρουσιάστηκε η έκθεση του κυρίου Καντέκ τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο η πρώτη παγκόσμια αγορά από πλευράς ε, προϊόντων αλληλείας αλλά εξαρτόμαστε κατά 65% από εισαγωγές. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας και να προβάλλουμε την αγορά μας σε σχέση με τις παγκόσμιες αγορές πέραν από τα ε, γενικά στοιχεία έχει και πιο συγκεκριμένα καθήκοντα το παρατήριο αυτό δηλαδή καταρχήν να εξασφαλίσει μία γρήγορη μετάδοση ε, καθημερινά ή εβδομαδιαία ε, διαθέσεως της τιμής σε όλους τους ενδιαφερόμενους με συγκεκριμένα, για συγκεκριμένα τουλάχιστον είδη ίσως όχι όλα και σε ορισμένα μέρη ε, ή σε ορισμένους ομολόγους μας όπως είναι η Νορβηγία και η Ισλανδία. Τέλος το παρατηρητήριο θα πρέπει να παρακολουθεί την ποσότητα και την τιμή ίσως όχι καθημερινά ή εβδομαδιαία αλλά μάλλον μηνιαία ή τριμηνιαία για το σύνολο της κοινοτικής παραγωγής και αυτό να το δούμε σε όλα τα στάδια του συστήματος και τέλος το παρατηρητήριο θα πρέπει να βελτιώσει τη γνώση μας και τονίζω το, τη γνώση μας και των δημοσίων οργανισμών κοινοτικών, εθνικών, περιφερειακών ή άλλων και ολόκληρου του τομέα σχετικά με την διαρθρωτική κατάσταση της αλίας και της υδατοκαλλιέργειας που εκεί ίσως θα χρειαστεί να ασχοληθούμε ετήσια για να δούμε ποιος παρουσιάζει τι και κάθε ε, και σε τι τιμή. Σήμερα το απόγευμα θα μπορούσαμε να επανέλθουμε στο Παγκάσιο που ήταν ενδιαφέρον. Ε, ή να δούμε πώς κατανέμονται οι εταιρείε ε, ή τα κέρδη σε όλες τις φάσεις αυτής της αλυσίδας. Και τέλος θα χρειαζόταν μία ανάλυση των τιμών, των πληροφοριών περί των τιμών, διότι αναφέρθηκα στη γέννηση αυτής της πρωτοβουλίας εις ε, την ανακοίνωση για την οικονομική κρίση και την κρίση των καυσίμων και στις δύο αυτές ανακοινώσεις πάντοτε ο τομέας ε, ε, ζήτησε να μπορέσει να επανακτήσει εντός της αλυσίδας τα κέρδη του διότι πίστευε ή μάλλον ε, διατηνόμενος ότι είχαν ε, ανισότητες όσον αφορά την υπόλοιπη ε, αλυσίδα και να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας στον τομέα αυτό. Τρίτον, πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Ίσως γρήγορα γρήγορα πρέπει να πω ότι καταρχήν το παρατηρητήριο αυτό θα πρέπει να συγκεντρώσει δεδομένα όχι να κάνει δηλαδή τάμπουλα ράζα, ε, θα εργαστούμε βάσει του ότι ήδη υπάρχει. Αλλά από τις πηγές αυτές θα πρέπει να συγκεντρώσουμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και να τις βάλουμε σε ένα κοινό κορβανά και σε μία δεύτερη φάση το παρατηρητήριο αυτό θα αναλάβει την επεξεργασία των δεδομένων δηλαδή να μπορέσει πραγματικά να τα επεξεργαστεί όπως είπα αφού τα συγκεντρώσει για να μπορέσει να παράγει ορισμένα υποπροϊόντα. Και τρίτον θα πρέπει να αναλύσουμε τα δεδομένα και η ανάλυση αυτή των δεδομένων θα επιτρέψει να παρακολουθήσουμε χρονικά τις εξελίξεις και ε, θα βασιστεί σε ορισμένες παραμέτρους που είναι βασικές για να βελτιωθούν οι γνώσεις μας και θα αναφερθώ σε ορισμένα από αυτά όπως παραδείγματο χάρη όπως είπα η εξέλιξη των τιμών στις ε, διάφορες φάσεις της αλυσίδας όσον αφορά το περιβάλλον ή το, ε, τα μακροοικονομικά συμφραζόμενα που θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε πού εξελίσσεται η αγορά αλίας και η εφόσον εξαρτώμαστε πάρα πολύ από εισαγωγές. Παραδείγματο χάρη έχουν σημασία και ισοτιμίε των νομισμάτων με τα οποία πληρώνονται τα προϊόντα αλληλεία, οι τιμέ των καυσίμων που επηρεάζουν πάρα πολύ ε, τις επιχειρήσεις και καινοτόμες αρχές σχετικά με τις ε, ε, ανάγκες των νοικοκυριών όσον αφορά τα προϊόντα αλληλεία και τέλος το παρατηρητήριο αυτό θα μπορέσει να διαθέσει αναλύσεις όσο δυνατόν σε περισσότερες κοινοτικές γλώσσες κατά τρόπον ώστε οι ενδιαφερόμενοι, τα κράτη και οι περιφερειακές αρχές να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για πολιτικούς στόχους τα στοιχεία αυτά. Τέλος ε, να σας πω γρήγορα πού βρισκόμαστε και ε, πού θα κατευθυνθούμε το πρόγραμμα έχει τρεις φάσεις. Η πρώτη είναι μια φάση διαπίστωσης, διαπιστώσεων, η οποία άρχισε το Φεβρουάριο και θα λήξει τέλη Ιουνίου. Είναι μια φάση κατά την οποία ο ετών θα πρέπει να ορίσει όλες τις πηγές δεδομένων που προϋπάρχουν και να εκτιμήσει την ποιότητα και την διαθεσιμότητα. Δεύτερο στοιχείο, ο ετών, ο συμβουλευόμενος, θα πρέπει να προτείνει λύσεις για την πλήρωση των κενών ως προς ε, ύπαρξη δεδομένων. Δηλαδή, ε, όλα τα δεδομένα στον, ε, σε επίπεδο που αφορούν το τομέα της αλίας. Αυτή η φάση θα λήξει τον Ιούλιο. Η δεύτερη, που θα χρειαστεί περίπου ένα χρόνο, θα αρχίσει στην αρχή του επομένου έτους και αυτή η φάση θα είναι μία ε, φάση σύλληψης και εκτέλεσης ως προς τα προϊόντα αλίας και υδατοκαλλιέργειας. Σε αυτή τη φάση ο συμβουλευόμενος με βάση τα δεδομένα και τις επισκέψεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διερευνήσει τις πηγές δεδομένων και τον ορισμό της προσπελασιμότητας της ε, πληροφορίες που θα τον απασχολήσουν. Το δεύτερο στοιχείο είναι να δούμε τι μπορεί να ε, δοθεί ως παραγωγή που θα ορίσει το παρατηρητήριο με γραφήματα, με ε, μνημόνια και ούτω καθεξής, ανάλογα με την περιοδικότητα παραγωγής. Η δεύτερη φάση σύλληψης παραγωγής αφορά το, την ε, αναγνώριση όλων των μέσων, υλικών και ανθρωπίνων για να λειτουργήσει αυτό το παρατηρητήριο καθώς και προτάσεις για τον τρόπο λειτουργίας, πώς αυτά τα νέα μέσα θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή. Και τελευταίο σημείο είναι να διασφαλιστεί ένα πληροφορικό μέσο στο ύψος των περιστάσεων. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε ένα πληροφορικό μέσο αρκετά περίπλοκο αλλά και αποτελεσματικό αν θέλουμε να ε, πετύχουμε τους διάφορους στόχους που σας προανέφερα. Με τη λήξη αυτής της φάσης, στα τέλη του 2011, μπαίνουμε στην τρίτη φάση που απαιτείται σε τέτοιες αποστολές. Είναι μια φάση δοκιμών και μεταφοράς. Διότι από την πείρα μας και με βάση την πείρα συναδέλφων από άλλους ε, τομείς, στο μέτρο της ε, γεωργίας, όπου υπάρχει παρατηρητήριο, τονίζουμε την ανάγκη αυτής της φάσης δοκιμών και μεταφοράς. Θα χρειαστεί μεταξύ 6 και 7 μηνών και θα λάβει χώρα το 2012, έτσι ώστε το παρατηρητήριο αυτό να είναι ένα ε, μέσον που να είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Αυτά είναι τα σημεία που ήθελα να θίξω για να σας περιγράψω αυτό το εγχείρημα και θα ήθελα εν κατακλείδη να επιμείνω σε τρία σημεία. Πρώτον, αυτό το μέσον δεν θέλει να ε, καταστρέψει όλα τα προηγούμενα, ούτε να τα αντικαταστήσει, αλλά με βάση των μέσων που προϋπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη να προσπαθήσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή ένα κοινοτικό μέσο για να βελτιώσουμε τις γνώσεις στον τομέα, τους διαφόρους ε, ε τομείς και υπευθύνους των, ε, των τομέων παραγωγής. Δεύτερον, θα ήθελα εντάχει να μιλήσω για τα δύο μεγάλα ραντεβού μας μαζί σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πρώτο είναι στη λήξη της πρώτης φάσης μετά από αυτή την αξιολόγηση και θα πρέπει και θα πρέπει να ξαναβρεθούμε κατά το τέλος του έτους για να σας ε, δώσουμε αυτή την πρώτη αξιολόγηση μετά από την έκθεση που θα υποβληθεί κατά τα τέλη Ιουλίου. Και στα τέλη του 2011 θα έχουμε το δεύτερο, τη δεύτερη συνάντησή μας γιατί μιλάμε για την κοινή πολιτική αλίας. Εάν αυτό το μέσο είναι αναγκαίο για την αναζωογόνηση της κοινής πολιτικής αλληλείας, θα πρέπει να εξευρεθεί μία ε, νομική βάση με βάση την κοινή πολιτική αλίας στο 2011. Ακόμα κι αν δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το μέσο, ήδη από το 2011 θα γίνει μία ε, συνάντηση και συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, Νομίζω ότι το παρατηρητήριο αυτό συστάθηκε μετά από επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλου του τομέα παραγωγής, του βιομηχανικού τομέα και επειδή προβλέπεται η πρώτη συνάντηση στο τέλος του έτους, θα είμαι στην διάθεσή σας να σας δώσω όσες πληροφορίες θέλετε και αυτό μπορεί να γίνει και σήμερα, αν το κρίνετε σκόπιμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάρτογκ από την ΕΠΗ θέλει να λάβει επίσης το λόγο, αν δεν κάνω λάθος. Πρόκειται για ένα διαφορετικό θέμα. Πρόκειται για την ενία θαλάσσια πολιτική. Άμα θέλετε μπορείτε να κάνετε την παρουσίασή σας και μετά θα μιλήσουν τα μέλη. Επειδή θα μιλήσω για δεύτερη φορά θα είμαι σύντομος γιατί ε, ασχοληθήκαμε με αυτό το ε, θέμα και στην προηγούμενη θητεία. Θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι η ενιαία θαλάσσια πολιτική δεν αντικαθιστά τους επιμέρους τομείς. Θέλουμε οι διάφοροι τομείς να έχουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Έχετε τέσσερα έγγραφα. Το έγγραφο προόδου, την ανακοίνωση για τη Μεσόγειο την εξω... και την εξωτερική διάσταση. Άρα τα χρήματα και η πολιτική συμβαδίζουν όπως θα σας ε, επεξηγήσω. Και αναμένουμε την έκθεση της κυρίας Μάισνερ για τα τέσσερα αυτά έγγραφα. Ως προς την ε, εκτέλεση του προϋπολογισμού νομίζω ότι τα καταφέραμε πολύ καλά. Οι πιστώσεις υποχρεώσεων ήταν 99,7% στον τομέα των δεσμεύσεων υποχρεώσεων. Για τα πιλωτικά είχαμε ένα 95%. Αλλά αυτό γιατί διαπραγματευτήκαμε πολύ καλά και δεν χρησιμοποιήσαμε τα υπόλοιπα χρήματα, δεν χρειαζόμασταν καν μας, αρκούσαν το, μας αρκούσε το 95% στις πιστώσεις πληρωμών λίγο χαμηλότερα τα ποσοστά διότι η εφαρμογή των μελετών χρειάστηκε περισσότερο χρόνο και ορισμένες πληρωμές του παρελθόντος έτους δεν έγιναν. Γι' αυτό έχουμε επίπεδο εκτέλεση 78% για προπαρασκευαστικέ και 65% για τα πιλωτικά σχέδια. Αλλά τα χρήματα αυτά θα δαπανηθούν αργότερα. Τώρα, τα χρήματα πού πηγαίνουν. Θα σας δώσω δύο ποσοστιαίες αναλογίες ως προς το συνολικό προϋπολογισμό, όχι μόνο για το 2009, αλλά 2007, 2008 και 2009. Ε, δεσμεύσαμε 20 εκατομμύρια και εν τρίτον πήγε στη, στη γνώση της θάλασσας, το 1 τρίτο, στην εποπτεία της θάλασσας και το υπόλοιπο στην εξωτερική διάσταση, μελέτες και βιώσιμα σχέδια. Πέρυσι σας μίλησα για το, την προσδοκόμενη έκβαση τι αναμένουμε στο τέλος. Βαθμιαία βλέπουμε ένα output ε, ως προς τη γνώση της θάλασσας. Τα, οι μελέτες θα οδηγήσουν στην πρώτη έκθεση προόδου τον Ιούνιο για να δούμε ποιες ε, γνώσεις, τι νέες γνώσεις υπάρχουν. Επίσης είχαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την εποπτεία της θάλασσας όπου συμμετείχε και η ακτοπλοεία για ελέγχους της θάλασσας από ε, διάφορα κράτη-μέλη, ένα εγχείρημα που στέφτηκε από επιτυχία. Οι Γάλλοι και οι Σουηδοί συμμετείχαν στα δύο αυτά προγράμματα. Έχει επιτελεστεί πρόοδος και αυτό το αναφέρω γιατί όταν η Επίτροπος Δαμανάκη ήρθε ε, εδώ στην ομάδα και μίλησε για τον Άτλαντα των θαλασσών. Ε, μας είπε ότι θα προωθηθεί σύντομα. Την επόμενη εβδομάδα θα ε, εκινήσουμε τη διαδικασία Άτλαντα των θαλασσών και θα ήταν κρίμα να μην σας έχω ενημερώσει για αυτό το, το περιορισμένο αλλά επιτυχές σχέδιο. Ο κύριος Γκάλαχερ ρώτησε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Το μέλλον βρίσκεται στα χέρια του νομοθέτη και της αρχής του προϋπολογισμού. Η Επίτροπος Δαμανάκη θα υποβάλει μία πρόταση που ενεκρίθη από την Επιτροπή για χαμηλές δαπάνες σε αυτόν τον τομέα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ευεργετηθούμε από τις δυνατότητες που μας ε, δίνει το Κοινοβούλιο για να παγιοποιήσουμε και να προωθήσουμε τις προσπάθειες που καταβάλαμε στους διάφορους τομείς. Αυτά εν είδη εισαγωγή, Πρόεδρε. Ωραία. Ευχαριστούμε και τον κύριο Χάρτοκ και τον κύριο Ραμπό από την Επίτροπη. Πρόκειται για ένα θέμα του προπολογισμού. Κυρία Ρόντας, θα θέλατε να μιλήσετε για κάποιο τμήμα αυτού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όχι για το τελευταίο θέμα, διότι νομίζω ότι εκεί είμαστε σε καλό δρόμο και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και τα δημοσιονομικά δημοσιονομικά μέτρα διαθέσιμα παρόλο που τελειώνει η τριετία τώρα και το ερώτημα είναι τι θα γίνει στη συνέχεια και από ποια γραμμή του προπολογισμού θα διετίθενται τα χρήματα. Αλλά είπατε ότι είσαστε καλά προετοιμασμένοι και φαντάζομαι ότι θα μπορέσετε να μου απαντήσετε γρήγορα. Αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι το παρατηρητήριο. Και θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ κάθε επιτυχία. Ε, με ενθουσίασαν οι οι ε, πληροφορίες ε, ε, έχουν συμμετάσχει και οι αλληλείς δέχτηκαν τα μέτρα αυτά γιατί εγώ εργάζομαι στη Γεωργία και ξέρω ότι παρόλες τις αρχικές κριτικές των Γεωργών τώρα υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός οπότε πιστεύω ότι ο στόχος αυτός είναι αξιέπαινος. Για τους στόχους αυτούς υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση στον προϋπολογισμό. Θα μπορέσουν να διατεθούν, θα επαρκέσουν ή θα πρέπει ε, στην ε, ε, νέα στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αλίας να προσθέσουμε πόρους. Είναι κάτι το οποίο οποίο θα ε, συζητούμε και με άλλους, αλλά αν μας πείτε ότι είσαστε έτοιμος θα είμαι πολύ ευτυχής. Ε, πριν από τον κύριο Ράμπο, ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σημερίζουν τι απόψει κυρία ρόντου κυρίως για ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό που είναι η δημιουργία αυτού του κέντρου για τη συλλογή των πληροφοριών. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή το εξή. Έχετε σκεφτεί να δημιουργήσετε πιο θετικά ε, μέσα από αυτά τα οποία χρησιμοποιεί η Eurostat. Διότι η Eurostat προς το παρόν δεν επαρκεί από ό,τι ξέρουμε, αλλά βεβαίως όλα εξαρτώνται από το χρόνο. Γενικά οι πληροφορίες φτάνουν αργά. Και η αξιολόγηση της Eurostat είναι μια αξιολόγηση που δεν μπορεί πάντα να αναλυθεί με λεπτομέρειες για να ξέρουμε γιατί ήδη μιλούμε όσον αφορά τις εισαγωγές τις εξαγωγές. Είπατε ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο κέντρο στο οποίο θα μελετώνται μόνο κάποια είδη. Υποθέτουμε λοιπόν λοιπόν, μπορούμε να υποθέσουμε λοιπόν ότι θα μελετηθούν ευθύ εξ αρχή μόνο κάποια είδη ή όλα τα είδη τα οποία μπορούμε να βρούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι άλλο. Μπορώ να υποθέσω ότι θα κάνετε μόνο ε, δουλειά για να βοηθήσετε κάποιους άλλους ή θα αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες και σε άλλα θέματα όπως φερειπίν αυτό της επίλυσης των διαφορών διότι στα πλαίσια της κοινή αλληλευτικής πολιτικής ή της υδατοκαλλιέργειας παρατηρούμε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες και αυτό είναι θεωρητικό παράδειγμα το οποίο σας δίδω τώρα δεν συμμορφώνεται με την κοινοτική αλληλευτική πολιτική και εισάγει πολύ μεγάλες ποσότητες του περίφημου παγκάσιου με πολύ χαμηλότερη τιμή από αυτή που κυκλοφορεί στην αγορά. Αυτό λοιπόν το νέο μέσο που θα έχετε, εκτός από το να κάνει αναφορές για το τι συμβαίνει ή να κάνει ε, εκτιμής και μελέτες θα έχει κάποιο είδους ε, νομική ισχύ ώστε να καταγγέλει την να γνωστοποιεί τέτοιου είδους ε, ε καταστάσεις. Ευχαριστώ κύριε Ράμπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο ερώτημα για τους αλείς. Ναι, δύο φορές λέω. Πρώτα απ' όλα, διότι ετήσι τους δημιουργήθηκε αυτή, το αυτό το μέσον και λύθη αυτή η πρωτοβουλία, πράγμα το οποίο άρχισε ως διαδικασία από την προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου, διότι εκφράσατε την βούλησή σας να δημιουργηθεί αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, αυτή η προπαρασκευαστική δράση, στην οποία δώσετε 4 εκατομμύρια. Δεύτερον, κάθε φορά που περνάμε στο επόμενο στάδιο, όλοι οι εκπρόσωποι του τομέα αυτού ενημερώνονται. Βεβαίως δεν ερχόμαστε σε επαφή με κάθε ελία χωριστά, αλλά με τους εκπροσώπους της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πρόοδο των εργασιών μας. Δύο φορές λοιπόν λέω ναι. Τώρα, αν αυτό αποτελεί λύση για τους αλληλείς, ναι, ε, συλλογικά αν θέλετε, διότι ο στόχος είναι να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας. Τις ε, οικονομικές γνώσεις που πρέπει να έχουμε στον τομέα αυτό. Και όλες αυτές τις γνώσεις να τις μεταφέρουμε και στους αλληλείς. Διότι κάποιες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες για τους αλληλείς και τη στιγμή την οποία επιθυμούν να βρουν αγορές για τα προϊόντα τους, θα μπορούν να έχουν πληροφορίες πιο λεπτομερείς και επικαιροποιημένε για τις αγορές τις οποίες ενδεχομένως θα ήθελαν να έχουν πρόσβαση για τα προϊόντα τους. Τώρα, αν υπάρχουν συμπληρωματικά κονδύλια, διπλή απάντηση θα σας δώσω. Κατά πρώτο λόγο, όχι, δεν χρειαζόμαστε για αυτή την δράση της, την προπαρασκευαστική συμπληρωματικά κονδύλια. Βεβαίως όμως είναι σαφές ότι αν στο τέλος αυτής της προπαρασκευαστικής φάσης μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα βιώσιμο σχέδιο το οποίο να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τις οποίες προανέφερα στους γενικούς και ειδικούς στόχους ανάλογα με την μορφή την οποία θα δώσουμε σε αυτό το παρατηρητήριο προβλέπεται ενδεχομένω να ζητήσουμε οικονομική υποστήριξη η ε, συγχρηματοδότηση από τον κοινοτικό προπολογισμό για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Άρα η απάντησή μου είναι όχι για να φέρουμε σε πέρα στο πιλωτικό μας σχέδιο μέχρι το τέλος του 2011 και θα δούμε μετά ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα προκαλέσει αυτή η προπαρασκευαστική μας δράση σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Τώρα, εάν αυτό το μέσον θα είναι καλύτερο από το ευρωμαρόμετρο. Βεβαίω είναι η απάντηση. Είναι καταφατική η απάντησή μα. Καταφατική διότι θα πρόκειται για κάτι το οποίο είναι εξειδικευμένο για τα προϊόντα αλληλεία και την καλλιέργεια. Έχουμε να κάνουμε εδώ με μια πάρα πολύ πολύπλοκη αγορά που αποτελείται από εκατοντάδε προϊόντα τα οποία έχουν, ε, παρουσιάζονται πολύ διαφορετικά τα μεν από τα δε και έχουμε πολύ διαφορετικές αγορές και εμείς θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο να ανταποκρίνεται σε αυτές τις αγορές. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα κάνουμε τα πράγματα πολύ καλύτερα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιδρούμε και πιο έγκαιρα, διότι τα δεδομένα που έχουμε σήμερα δεν είναι πολύ ενδιαφέροντα για το σύνολο του κλάδου και πολλές φορές θεσμικά όργανα που πρέπει να πάρουν αποφάσεις δεν έχουν ε, ε, διάθεσή τους για τον τομέα της το και της ελίας ενημερωμένα οικονομικά ή άλλα στοιχεία. Με ρωτήσατε αν ο στόχος είναι να περιοριστούμε σε κάποια είδη. Εξήγησα ότι είναι πολλαπλό ο στόχο μα. Όταν έχουμε πληροφορίες πολύ συγκεκριμένες, τι οποίε χρειαζόμαστε για να πάρουμε μια απόφαση οικονομική και όχι απαραίτητο οικονομική, θα μπορούσαμε να το κάνουμε βασιζόμενοι σε κάποια είδη τα οποία θα έχουν επιλεγεί ως αντιπροσωπευτικά για να μας πούνε βραχυπρόθεσμα ποιες είναι οι τάσεις. Αυτό δεν μας εμποδίζει βεβαίως να έχουμε στη διάθεσή μας όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για άλλα προϊόντα. Θα συλλέξουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά για κάποια προϊόντα ή για κάποιους στόχους θα επιλέξουμε κάποια προϊόντα. Και εδώ το σημαντικό ερώτημα που τίθεται είναι εάν ο τελικός στόχος του παρατηρητηρίου είναι να έχουμε ένα επικουρικό μέσον για να λαμβάνουμε αποφάσεις και για να βοηθούμε τον επαγγελματικό αυτό κλάδο ή εάν το παρατηρητήριο αυτό θα είναι σε θέση να παίρνει μέτρα και να λαμβάνει κυρώσεις κατά αυτών οι οποίοι δεν τηρούν. Τι δεν τηρούν? Τους κανόνες. Ποιους κανόνες που έχουν ε, θέσει άλλοι. Ναι, όντως πρόκειται για υποστηρικτικό παρατηρητήριο. Υποστηρίζουμε τις δημόσιες αρχές που έχουν πολιτικές υποχρεώσεις, αλλά όντως πρόκειται και για ένα μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας και στη διάθεση όλων ασχολούνται με την αλία. Από, την, από τον παραγωγό, τον αλιαία, μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Αυτά ήθελα να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε, σε ερωτήσεις που μου τέθηκαν. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, πρόκειται για προτάσεις οι οποίες προήλθαν από την δική μας αλληλευτική επιτροπή στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό το λόγο ήταν καλό που μας έδωσε, ε, μας έκανε αυτή την ενημέρωση η Επιτροπή για να μας πει και σε θέματα προπολογισμού πώς μεταφράζονται οι προτάσεις που κάναμε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε ε, Γαμπό, κύριε Χάρτογκ για αυτές τις προφορίες που μας δώσατε και θα σας ξανακούσουμε όταν θα ολοκληρωθούν τα σχέδια με τα οποία ασχολείστε. Λοιπόν, στην αρχή της σημερινή μας συνεδρίαση σημείωσα ότι δεδομένου ότι είχαμε προβλέψει ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο στη δεσίμα σήμερα το απόγευμα και μετά από μία πρόταση που είχαμε από την, ε, το τμήμα πολιτικής για θέματα συνοχής, καλέσαμε τον συντάκτη της έκθεσης. Έχει σημασία το μέγεθος μέσα για την διαχείριση των ολιευτικών στόλων. Την έκθεση αυτή την συνέταξε ο κύριος Βανχόφ, ο οποίος μας παρακολούθησε μεγάλη υπομονή όλη την ημέρα συνεδριάσης μας. Κύριε Βανχόφ, σας παρακαλούμε τώρα να κάνετε μία παρουσίαση του θέματός σας και στο ίντερνετ. Έχετε το λόγο κύριε Βανχόφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Ευχαριστώ μέλη της Επιτροπής Ελίας. Θα σας ευχαριστήσω όλους τους παρόντες στην αίθουσα και στην ερώτηση, η ερώτηση που τίθεται πολύ συχνά είναι έχει σημασία το μέγεθος και νομίζω ότι αυτό στον, για τον ελληνικό στόλο είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Θα προσπαθήσω σήμερα το απόγευμα να σας πω βασικά γιατί μας ανατέθηκε αυτή η μελέτη, τι κάναμε στα πλαίσια αυτής της μελέτης και πριν να προχωρήσουμε θα σας πω πώς μπορούμε πρώτα απ' όλα να ορίσουμε την ε, ε, δυνατότητα αλίευσης, πώς την μετρούμε, πώς την ορίζουμε και πώς την ε, διαχειριζόμαστε. Ο στόχος μας ποιος είναι. Αρχίσαμε βασικά με μία δημοσίευση του, της ΕΦΑΟ του 1999 για το Διεθνές Σχέδιο Δράσης για την διαχείριση της ε, δυνατότητας και αλίας. Εάν εξετάσει κανείς την πράσινη βίβλο της κοινής, της, για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής θα δείτε ότι υπάρχει ακόμη υπεραλίευση εκ μέρους των ε, αλληλευτικών του κοινοτικού στόχου και αυτό είναι πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Μου ζήτησε η υπηρεσία πολιτικής να δούμε τα συστήματα διαχείρισης της Αλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και των ΗΠΑ. Και να δω κατά πόσον θα μπορούσαμε να μάθουμε από τις δικές τους εμπειρίες και να δούμε αν θα μπορούσαμε στο πλαίσιο της Ευρώπης να εφαρμόσουμε ένα παρεμφερές σύστημα διαχείρισης. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ορίσουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για δυνατότητες αλίας είναι, αφορά το ποσοστό ε, των αλλιευμάτων που μπορεί κανείς να αλλιεύσει. Πριν να συζητήσουμε την υπεραλίευση θα πρέπει να κάνουμε διαφοροποίηση μεταξύ πλεονασματικής δυνατότητας αλίευσης και υπεραλίευσης. Υπάρχει διαφοροποίηση. Η Ε, σε σχέση με το παρόν επίπεδο αλίευσης έχουμε ένα συμπληρωματικό ε, ποσό σε σχέση με το σύνελο επιτροπωμένων αλίευματών για κάποια χρονική περίοδο ή μιλάμε και εδώ έχουμε να κάνουμε excess capacity ή για over capacity που είναι η υπεραλίευση όπως λέμε στα ελληνικά. Κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι η διαφοροποίηση μεταξύ της ανάλυσης που αφορά το input και αυτής που αφορά το output. Στην πρώτη περίπτωση το input είναι πόσα αλλιεύματα μπορούμε να αλλιεύσουμε με τον παρόντα στόλο που διαθέτουμε. Η output ανάλυση είναι αυτή η οποία αφορά το πόσα πόση αλλιευτική δυνατότητα πρέπει να έχουμε για να επιτύχουμε το ανώτατο όριο του συνόλου επιτρεπωμένων αλλιευμάτων. Λοιπόν, ας μετρήσουμε την δυνατότητα της ε, ικανότητας αλλιεύσης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την αλλιεύση, με τον στόλο και, το 2000, και με άλλες ιδιαιτερότητες. Το 2007 στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι όντως για πολλά χρόνια χρησιμοποιούμε την, ε, το τονάζ των λευτικών στόλων και την δυναμικότητα των μηχανημάτων για να κάνουμε κάποιες μετρήσεις. Αυτός είναι ένας ε, πολύ σημαντικός δείκτης που χρησιμοποιούσαμε τότε και φανταστείτε αν έπρεπε κανείς να μετρήσει τις στράτες που κάνουν ε, την ε, αλίευση πελαγικών και μη πελαγικών ειδών, σε τι ε, συμπεράσματα θα καταλήγατε αν κάνατε αναφορά μόνο στα δυναμικότητα του κάθε μηχανήματος. Διότι οι τράτες φερρυπίν δεν έχουν πολύ δυνατότητα, έχουν χώρο πιάνει το μηχάνημα και δεν έχουν μεγάλη δυνατότητα ε, αποθήκευσης. Επίσης, είπαμε ότι θα πρέπει να μετρήσουμε πώς θα μπορούσαμε μετρώντας την ε, δυναμικότητα της μηχανής και τα δίχτυα να κάνουμε διαφοροποίηση της μέτρησης. Τις διάφορες ανακοινώσεις επιτρεπηθείς για μεγάλες κατηγορίες χρησιμοποιεί τα διάφορα είδη αλευτικών σκαφών όπως οι τράτες ή άλλα είδη μηχανοκίνητων αλευτικών σκαφών για να κάνει κάποιες μετρήσεις. Παραγάδια και τα λοιπά. Τέτοια διαφορετικά είδη. Ε, ανάλογα με την μηχανή, είπαμε, του αλευτικού σκάφους. Και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη. Κάτι άλλο το οποίο πρέπει να αναφέρω είναι η δουλειά που κάνει η Τεχνική και Επιστημονική Επιτροπή που βοηθά την Κομισιόν στη δουλειά της για την θέσπιση της ε, ε, πολιτικής αλίας και πριν από τέσσερα χρόνια δημοσιεύθηκε μια έκθεση για την διαθέσιμη δυνατότητα αλίευσης και την διαθέσιμες ε, ευκαιρίες αλίευσης δεν μπόρεσε να γίνει συγκριτική ανάλυση δεδομένου ότι υπήρχε έλλειψη δεδομένων. Ξέρουμε ότι στα πλαίσια των στατιστικών έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Στην αίσθηση ECF όμως, στην Επιτροπή αυτή είπαμε πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε δείκτες για να ξέρουμε ποια είναι επί τόπου κάθε φορά και ανα πάσα στιγμή η ισορροπία που υπάρχει μεταξύ της δυνατότητας αλίευσης και των ευκαιριών αλίευσης. An Επίσης, είπαμε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται και άλλοι κοινωνικού ή βιολογικού περιεχομένου δείκτες και όχι μόνο οικονομικοί. Και πάλι, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά βλέπετε εδώ ότι είναι δυνατόν από τον οικονομικό ε, τομέα, από τον βιολογικό και από τον κοινωνικό να έχουμε διάφορους δείκτες του οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, βιολογικοί δείκτες. Τι εξετάζουν. Την θνησιμότητα των αλλιευμάτων και την ε, προσπάθεια αναλλιευόμενη ομάδα. Επίσης, έχουμε όπως σας είπα, τις ε, μελέτες της Κομισιόν και της ειδική αυτής τεχνικής επιτροπής για να μπορέσουμε να μετρήσουμε όλους αυτούς τους δείκτες. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι η δυνατότητα αλίευσης είναι κάτι το οποίο πολλές φορές δεν είναι πολύ σημαντικό. Εξαρτάται για τι είδους δυνατότητα μιλάτε. Στον τομέα των αυτοκινήτων ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτοκίνητα με ε, ανάπτυξη ταχύτητα διαφορετική, μικρή, μεγάλη. Αν θέσετε όμως ανώτατο όριο έχει λυθεί το πρόβλημά σας. Από οικονομικής πλευράς όμως, εδώ έχουμε να κάνουμε ε, με αν λάβουμε υπόψη τον οικονομικό δείκτη, με πλοία των οποίων οι δυνατότητε αν θέσουμε τέτοιου οικονομικού στόχου πάνε χαμένες. Τώρα, για να διαχειριστούμε την ε, ε δυνατότητα αλίευση, μπορεί να έχετε. Και για να διαχειριστείτε το όλο θέμα, ή ε, κανονισμούς που να διευθετούν τα αλλιευόμενα ε, είδη ή να έχετε κανονισμούς που να διευθετούν το κάθε αλίευμα ή να έχετε οικονομικά μέτρα που διευθετούν την συμπεριφορά και τις προσαρμογές των αλλιέων όταν ασκούν αυτή τη δραστηριότητά τους. Έχετε εδώ ένα πίνακα στον οποίο έχετε έλεγχο του input, έλεγχο του output, διάφορες αλλαγές, έχετε τα μέσα που χρησιμοποιούνται και τις χώρες οι οποίες ε, χρησιμοποιούν τα διαφορετικά μέσα τα οποία διαθέτουμε. Εμείς και όλος ο κόσμος. Στην Αυστραλία χρησιμοποιείται ένα σχήμα αναγωγής σε μονάδα όλων των μετρήσεων. Δηλαδή κάθε φορά μελετάτε το μέγεθος της μηχανής και του ε, αλληλευτικού σκάφους δίδονται κάποιοι βαθμοί, κάποιες μονάδες και μετά αυξάνονται, αφαιρούνται, προστίθενται και γίνονται κάποιες μετρήσεις. Στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Ισλανδία, στην Νορβηγία. Έχετε ε, διαφορετικού είδους μέσα που χρησιμοποιούνται. Ε, ποσοστώσεις μεταφοράς ε, επίσης ε, αλλιευτικών δραστηριοτήτων. Το πιο σαφές μέτρος είναι η διαχείριση του αριθμού αδειών αλίευσης που χορηγείται. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βρίσκουμε στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Ισλανδία, στην Νορβηγία, στην, στην Νορβηγία Στην, ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα μοναδικό στο είδο του ε, σχήμα εισόδου-εξόδου και επίσης στις Ηνωμένε Πολιτείες, στον Κανδά, στην Αυστραλία και στην Νορβηγία έχετε το θέμα της καταστροφής των κάποιων περχαιωμένων λευτικών σκαφών και το θέμα των αδειών τα τάξ, τα περίφημα σύνολο επιτροπωμένου αλλιεύματος τα έχετε στην... Ε, also familiar with all the, uh, Έχετε το θέμα επίση τώρα στο, στον έλεγχο του output, τα τάξ, τις ποσοστώσεις, τις ατομικές ποσοστώσεις που δίδονται στις, ε, στους συνεταιρισμούς, ε, στις διάφορες κοινότητες, σε προγράμματα περιφερειακά, σε σύνολο αλλιευτικών σκαφών, μεταφορά ποσοστώσεων και δικαιώματα αλλίευσης, όπως τον Καναδά, την Αυστρία, την Νέα Ισλανδία, την Ισλανδία και διαχείριση ε, ανάκτησης κόστους στη Νέα Ζηλανδία και στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται λεπτομεριακά όλα αυτά τα στοιχεία, όλα αυτά τα μέσα. Δεν θα πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Νομίζω ότι θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια άλλα θέματα τώρα. Πρώτα απ' όλα, η διαχείριση της δυνατότητας που έχουμε για αλήψη είναι κάτι το οποίο θεωρείται σε όλες τις χώρες σαν προτεραιότητα ο Καναδάς, η ΙΠΑ και η Αυστραλία έχουν ειδικά ε, συστήματα αντιστάθμισης buyback σχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για να εάν θέλει κανείς να μειώσει την δυνατότητα αλίευσης. Γιατί αν δεν δώσουμε κάποια αντισταθμίδα, σε μερικά χρόνια θα ξανακαταλήξουμε στην ίδια κατάσταση, εάν προτείνεται να μειωθεί η δυνατότητα αλίευσης. Τι βρίσκουμε σε διάφορε περιοχέ του κόσμου και κυρίω αν σκεφτούμε τη ΣΥΠΑ, που είναι μια τόσο μεγάλη χώρα, όπω και η Αυστραλία που έχει προηγμένε μεθόδου, έχετε διαφορετικές αλλιευτικές περιοχές και αλλιευτικούς στόλους και ειδικέ ρυθμίσεις που αφορούν ε, τοπικές πρακτικές, παραδοσιακά δικαιώματα και βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε διαφοροποίηση μεταξύ των διαφορετικών περιοχών και αλλιευτικών στόλων. Και το σημαντικό ερώτημα είναι τέτοιου είδους οι χρησιμοποίηση τέτοιων μέσων φέρουν αποτελέσματα. Δεν ξέρω τίποτε, διότι ο καθένας έχει το δικό του σύστημα αξιολόγησης των μέτρων που εφαρμόζει και βεβαίως κανένας δεν εφαρμόζει ένα μόνο μέτρο, πρόκειται για συνδυασμό. Και όπως σας είπα πριν από λίγα λεπτά όλα τα μέσα αφορούν την κάθε είδους αλληλεία και το κάθε είδους αλληλευτικό στόχο. ένα σύστημα λοιπόν που ισχύει για τη ΣΥΠΑ δεν μπορείτε να το αντιγράψετε για την Ευρώπη και να είστε σίγουρος ότι θα εφαρμοστεί με επιτυχία. Παρ' όλα αυτά, τι μπορούμε να δούμε σε όλες τις χώρες τις οποίες εξετάσαμε, ότι η δυνατότητα αλλιεύσης έχει μειωθεί τα τελευταία 10 με 15 χρόνια και φαίνεται ότι υπάρχει και η κοινή άποψη ότι η σημερινή ε, δυνατότητα, δυναμικότητα που προσφέρεται είναι πολύ μεγάλη. Κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις. Τα Τάξ είναι το κύριο, η κύρια αρχή στην οποία βασίζεται κανείς. Δηλαδή πρώτα πρέπει να καθορίζει ποιο είναι το σύνολο των επιτρεπομένων αλλιευμάτων. Και είδα επίσης ότι υπάρχουν, και αυτό με εξέπληξε, και ε, διαφορετικά συστήματα εξατομικεμένα συστήματα ποσοστώσεων. Τα ITQs, αυτά τα ατομικά ε, συστήματα ποσοστώσεων, αναπροσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τις δυνατότητες σε Αυτό τον λέγουν στην Ισλανδία ή στην Αυστραλία. Τώρα, από όλες αυτές τις εμπειρίες ποιο είναι το κύριο συμπέρασμα στο οποίο καταλέγουμε ότι βεβαίως όλα αυτά εξαρτώνται και από τις δυνατότητες που προσφέρει η αγορά. Έτσι λοιπόν ξαναφτάνω πάλι στο πρώτο μου ερώτημα. Η διάσταση, το μέγεθος έχει σημασία. Η υπεραλίευση δεν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει μόνο από οικονομικής πλευράς αλλά και από την πλευρά της διατήρησης. Με σωστό έλεγχο και εποπτεία των μέσων ε, που χρησιμοποιούνται για τους τόλους και τις δυνατότητες αλίευσης μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον από την Κομισιόν ως προς την αναθεώρηση της κοινή οργάνωσης της αγοράς, σκεφτόμαστε να εισαγάγουμε αυτά τα ITR και γνωρίζω στην Ισλανδία όταν συνέβη αυτό παγιοποίησε το καθεστώς, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αλλιών. έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε και τα πλεονάσματα. Και η Κομισιόν χαίρεται για την ύπαρξη αυτής της, αυτής της ιδέας, γιατί δεν χρειάζεται αντιστάθμιση. Όμως τα δικαιώματα αλίευσης παραμένουν στα χέρια πολύ ολίγων. Και αυτό σημαίνει ολοένα και λιγότεροι εργάζονται στον τομέα. Αυτό συνέβη στην Ισλανδία. Όταν μιλάμε για ITR, έχουμε σε αμηχανία. Ξέρω ότι το πλεόνασμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ίσως οι δυνάμεις της αγοράς είναι ένας μη δαπανηρός τρόπος για να καταφέρουμε κάτι τέτοιο. Θεωρεί η Ευρώπη ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις, ε, πλε, τις ε, πλεονασματικές ποσότητες. Θέλετε την προσωπική μου θέση, απάντηση, δεν έχω ιδέα. Αυτό που με εξέπληξε είναι ότι χρησιμοποίησαμε εμπορεύσιμα ή ανταλλάξιμα μέσα όπως τα ITQs. Τα ITQ, τα εμπορεύσιμα δικαιώματα, αγοράστηκαν από περιβαλλοντικές οργανώσεις και μετά αποδόθηκαν εκ νέου για να αλλιεύσουν υπό περιορισμούς. Ίσως αυτός είναι ένας τρόπος. Τα ψάρια ανήκουν σε όλους, άρα ο καθένας ε, θα πρέπει να έχει το μερίδιό του και να κάνει τι θέλει με αυτό. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν αλλιευτικοί στόλοι και υπάρχει ήδη ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Και με τη μείωση των ποσοστώσεων θα είναι πολύ πιο δύσκολο για αυτούς που θέλουν να παραμείνουν στην αγορά. Όμως από την καλή πλευρά ε, είχαμε χρηματοδότηση τομεακών προγραμμάτων. Εγώ προέρχομαι από την Ολλανδία, το καταλαβαίνετε και από την προφορά μου. Εάν ε, προσπαθήσουμε να διαβλέψουμε την πραγματικότητα είναι ότι, ότι αν βγάλουμε το ίμιση του αληφτικού στόλου, το άλλο ίμιση θα είναι πολύ υγιές. Βεβαίως αυτοί που παραμένουν θα πρέπει να καταβάλουν το τίμημα αυτών που αποχωρούν. Τι πρέπει να κάνουμε για την ε, υπεραλίευση. Άμα δω ε, τη, το δικό μας στόλο, ξέρω ότι μπορεί να απαλληφθεί μελλοντικά. Όμως εάν οι βιολόγοι έχουν δίκιο, θα ήταν κρίμα να έχουμε χάσει τον αλλιευτικό μας στόλο, αν έχουμε ανάκτηση αλλιευμάτων. αλλά πώς μπορούμε να βρούμε τα κατάλληλα μέσα. And... Uh, Παραδείγματος χάρη για τους αλλιευτικούς στόλους ρέγκας που έχουμε εμείς, μπορεί κάποια στιγμή να φύγουν οι στόλοι από τη, μέσα, από τη μέση, αλλά να έχουμε ανάκτηση ποσοστώσεων αλλιευτικών ειδών όπως η ρέγγα. θα έχουν εφιάλτες οι αλείς όταν ακούν ότι ορισμένες μη κυβερνητικές αγοράζουν αυτά τα δικαιώματα και τα επανακατανέμουν. Ε, υπάρχουν πολύ πλούσιες μη κυβερνητικές που έχουν πολλά, πολύ περισσότερα χρήματα από τις αλλιευτικές επιχειρήσεις. Δηλαδή αγοράζουν αλλιευτικά δικαιώματα και μετά τα επαναπολούν. Ναι, άρα ακόμα περισσότεροι εφιάλτες. Υπάρχουν μέλη της Επιτροπής που θα ήθελαν να σχολιάσουν. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ό,τι και να κάνουμε δεν λύνουμε το πρόβλημα και καλό θα ήταν τώρα να ε, διερευνούμε με μεμονωμένες λύσεις προσωπικές διότι ένα από τα ε, επιστημονικά μας Ινστιτούτα που επισκέφτηκα την περασμένη εβδομάδα στη Γερμανία έχει αρχίσει και σκέφτεται εάν δεν θα ήταν καλό να αναθέσουμε μεγαλύτερες ευθύνες εις ε, τους αλείς και εγώ μπορώ να δεχτώ πολύ καλά αυτή την πρόταση Απ' την άλλη πλευρά είναι, υπάρχουν και προβλήματα. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας πολλά χρόνια και σαν επιχειρηματίας πρέπει να επιχειρώ. Χωρίς λοιπόν να είμαι προκλητική δεν μπορώ να ζητώ ένα κοινωνικό ταμείο. Δηλαδή κάθε επιχείρηση έχει μία κοινωνική ευθύνη και θα είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε ίσως περισσότεροι δηλαδή αν στην Αλία δεν πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν δημόσια αγαθά όπως και στη γεωργία στην γεωργική πολιτική ε, σκεφτόμαστε εάν η γεωργοί δεν είναι υποχρεωμένη ε, να ασχολούνται υπεύθυνα για την παροχή ορισμένων ε, ειδών δημοσίων εφόσον πληρώνονται και αυτό μπορεί να ισχύσει και για την αλληλεία κατά τρόπον ώστε να έχουν και οι αλληλείς κάποιο σταθερό εισόδημα είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε αλλά βεβαίως είναι γεγονός και ελέγχθη ότι αν θέλει κανείς ε, να ερμηνεύσει διαφορετικά ε, την ε, υπερβολική, το, υπερβολικό, το πλεονάζον δυναμικό του αλλιευτικού στόλου καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη ότι θα μειώσουμε τους κινδύνους στη θάλασσα ε, να, εάν πείσουμε τους αλληλείς να κατανοήσουν ότι υπάρχουν κίνδυνοι και εκεί ε, και υπάρχει υπερβολική, ε, υπερβολικά μεγάλο στόλος. Πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολλές λύσεις και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όποιος πάει γρήγορα δεν δημιουργεί τόσα πολλά ατυχήματα όσο αυτοί οι οποίοι καθυστερούν. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας η οποία συνάδει πολύ με την συζήτηση που είχαμε τώρα για την κοινή αλευτική ε, ε, πολιτική στα διάφορα σήμερα το πρωί ε, πριν από το, τη διακοπή για το μεσημέρι είχαμε θίξει το θέμα της πετρελοκυλίδας στον κόλπο του Μεξικού και στην επόμενη συνεδρίαση θα το συζητήσουμε σαν σημείο της ημερήσιας διάταξης με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 17 Μαΐου 5 ε, ε, με 7 θα συζητηθεί αυτό το θέμα, στο, θα συνεδριάσει η Επιτροπή μας στο Στρασβούργο. Θα ήθελα ένα θέμα να τεθεί στα πρακτικά. Κάθε χρόνο έχουμε στην, ε, στις Βρυξέλλες την έκθεση Seafood. Ε, θα έπρεπε σαν Επιτροπή και όχι μόνο σαν, επιχειρή, σαν μεμονωμένα άτομα να επισκεφθούμε την έκθεση αυτή διότι θα μπορούσαμε να διεξάγουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Εξαιρετική ιδέα. Νομίζω ότι η Επιτροπή υπό μαλά συνθήκες οργανώνει ε, να έχει ε, εισιτήρια προσκλήσεις ε, για να πηγαίνουν τα μέλη της Επιτροπής. Το να πάμε σαν αντιπροσωπεία έχω σκεφτεί και εγώ ότι σε εκθέσεις γεωργικές στα κράτη-μέλη υπάρχει κυβερνητική παρουσία με την αναθεώρηση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής που είναι τόσο ενδιαφέρουσα καλό δεν θα ήταν ε, του χρόνου να έχουμε και ένα στάντ, ε, ένα περίπτερο ε, ή μία θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου ο κάθε ένας θα μπορούσε να έρθει να μας προσεγγίσει και εξεναλλαγής στις τέσσερις ημέρες που κρατάει το seafood θα μπορούσαμε να έχουμε συνεχή εκπροσώπηση. Βέβαια εξαρτηθεί από το κόστος αλλά θα μπορούσαμε έτσι να απαντήσουμε και σε ε, ερωτήσεις σχετικά με την αναθεώρηση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής που μέχρι τότε θα έχει διαμορφωθεί. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους παριστάμενους που συμμετείχαν και ευχαριστώ και τους υπολείπους που ήρθαν εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους.